I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Κούν. Καλημέρα σας. Ερχόμαστε στη δεύτερη μα συνεδρία σε αυτή τη βδομάδα. Πρόκειται κυρίως για τις ψηφοφορίες, αλλά πρώτα να σας αναφέρω τα αποτελέσματα των, της συνεδρίασης των συντονιστών. Σας έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 12, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από εσάς. Ψηφοφορίες. Λευκή βίβλος για τις μεταφορές. Και εδώ θα πρέπει να ρωτήσω καταρχήν αν το ΕΛΚ θέλει να λάβει το λόγο. αν είσαστε επαρκείς, αν έχετε αρκετούς ε, βουλευτές καταρχήν ή όχι. Μόνο τρεις είσαστε. Λοιπόν, τελειώνει η δοκιμαστική ψηφοφορία, όλα είναι εντάξει. Εντάξει. Θα σας ελέγχουμε στη συνέχεια. Στην αρχή είναι εντάξει, αλλά μετά μπορεί να έχετε περισσότερους ή λιγότερους. Λοιπόν, το blog των... Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε και χωρίς κάρτα. Ξεκινάμε. Έχουμε λοιπόν τον μπλοκ των τροπολογιών συμβιβασμού. Βλέπετε ποιες δεν περιλαμβάνονται στο μπλοκ. Βλέπετε την ε, τροπολογία 1, η οποία πρέπει να ψηφιστεί χωριστά. Αυτές οι οποίες δεν έχουν αστερίσκο όμως, όπως στην περίπτωση της τροπολογίας 2, Συμβαστική τροπολογία 2 περιλαμβάνεται στο μπλοκ το οποίο ψηφίζουμε καταρχήν. Η πρώτη ψηφοφορία λοιπόν είναι για το μπλοκ των τροπολογιών συμβασμού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. 92 υπέρ κατά άποχες κάνουμε ε, έλεγχο ηλεκτρονικό άρχεται η ψηφοφορία ένας περισσεύει από το ΕΛΚ πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται 17-23. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 117 με προφορική τροποποίηση. Έχετε αντιρρήσει για την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 με 23 απορρίπτεται. Εκατόν Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μα είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εντάξει να ελέγξουμε όπως θέλετε αυτή την ψηφοφορία. Για την 119. Πάλι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Και από τους σοσιαλιστές περισσεύει ένας. Έχετε ένα παραπάνω, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26-16 εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. <clears throat> Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 140. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 5 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η έξι έχει ρυθμιστεί. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 208. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-24. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης έλεγχος. Ξεκινάμε. Για την 209. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάουλ, με ακούς. Άρχεται. Πέρας. 21-22 απορρίπτεται. Καλά που σκέφτηκα να κάνω έλεγχο. Γιατί και με ισοψηφία πάλι απορρίπτεται. 2-12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23-20 εγκρίνεται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 15.30. 2.51 <clears throat> υπέρ κατά χέρι Συγκρίνεται. 252 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 264 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 263 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 262 υπέρ α εκπίπτει συγγνώμη 266 υπέρ κατά αποχές δεκτή 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 275 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε 275 ελέγχουμε άρχεται Άρχεται είπαμε. Πέρασε. 17-28 απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίτη. 2-79, υπέρ. Κατά. Αποχές συγγραφέτε, 2-80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2-81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 282. Άρχεται. Πέρας. 19-24 απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.98. <clears throat> Άρχεται η ψηφοφορία λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται. Με σαφήνεια. 2.98 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε και αυτό. 2.98 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίπτη. 2.99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 300. Απορρίπτεται. 301 υπέρ. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. 301. Πέρας. 24-19 εγκρίνεται. Όχι. 304 <clears throat> πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 324 κατά αποχές εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε 319 έλεγχος άρχεται Πέρας. Εγκέκριται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.31 υπέρ κατά ελέγχουμε την 3.31 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 3.48 έλεγχος άρχεται την ψηφοφορία. Πέρασε. 19.23 απορρίφθηκε. 3.46 υπέρ Αποχές απορρίπτεται. 3.59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.60 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. 3.60 ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. 17-25 απορρίπτεται. 361 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 364 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος βεβαίως. 364 Άρχεται. Πέρας. Από ρίπτεται 1924. 360-365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 366 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 366 Άρχεται. Πέρασε. 20-23 απορρίπτεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 370. Α, ήταν η ίδια μαζί. 371 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 371. Άρχεται. Πέρας. 23-19 εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 387 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 388 <clears throat> υπέρ κατά να ελέγξουμε 388 άρχεται η ψηφοφορία τέρας ψηφοφορίας 20 με 23 απορρίπτεται η 2024 καλύτερα. Ερχόμαστε στην 394 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 395 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σύμβαστη 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ 408 κατά αποχές απορρίπτεται. 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 419 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φροχτηρίας. Απορρίπτεται. 4 23 υπέρ. Κατά. Αποχές πάλι θα ελέγξουμε. Δεν ψηφίζεται όλοι μάλλον. 423 λοιπόν άρχεται. Οι, οι σοσιαλιστές έχουν ένα που περισσεύει. Εντάξει τώρα. Πάλι ένας περιπλέον στους σοσιαλιστές. Πέρας. 21-21 απορρίπτεται. Αλλά έχουμε, τη... έχουμε τον uh, κύριο Χόγκς ο οποίος είναι υπέρ. 22-21 εγκρίνεται. Δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. 4-38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.54 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για την 4.54. Άρχεται. Τέρας. Απορρίπτεται. Και έχουν 14 αποχές εδώ όπως βλέπετε. 4.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, όχι, δεκτή, δεκτή, δεκτή, συγγνώμη. Θέλετε έλεγχο. Καλά. Ήταν σαφές, αλλά θα ελέγξουμε και πάλι την συμβαστική 29. Άρχεται. Πέρας. 28-15 κρίνεται. 4-65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4-57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 457 άρχεται. Πέρας. 22-20 εγκρίνεται. 460 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 470 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 469 και 467 και 260 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Εκπίτη 468, 476 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 490 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος. 4.90. Άρχεται. Πέρας. 22-21 Ρόμπερτ, υπέρ. 23-21, ωραία. 4.93, υπέρ. Κατά αποχές θα κάνουμε έλεγχο. 493. Άρχεται λοιπόν. 21.24 21-24 απορρίπτεται. 494 υπέρ κατά άποχες θα κάνουμε έλεγχο. Άρχεται. Πέρας. 20-23 απορρίφθηκε. 504 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχο στην 504. Άρχεται. 1924 19-24 <laughs> απορρίφθηκε. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κάνουμε ένα σάλτο τώρα και πηγαίνουμε στην Συμβαστική 32. Α, συγγνώμη, 31, 31 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.25 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε 6.25 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Για την 23. Πέρας. 20-23 απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32. Αφήνω να την ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. 13-19 εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά Απόχες να λέξουμε. Για την 47. Άρχεται. Πέρας. 23-19 εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Σαφές ήταν αλλά θα το ελέγξουμε στην 56 άρχιτε. Πέρας 23-19 23-20 καλύτερα 73 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 76. Άρχεται. Πέρας. 23-20 εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 και 3 μαζί. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 καθώς και 2 καθώς και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά α, ας ελέγξουμε την 7 άρχεται πέρας από 1924 <clears throat> τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Άρχεται είπα. Πέρας. 37 με έναντι 38, 3 με 5 αποχές ε, συν χαρητήρια κύριε Φανεκάμπ. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, η εισηγήτρια είναι η Χένα Βίρκουμεν. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα η τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 5, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 5. Άρχεται. Πέρας. 25 προς 18 εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές ε, πρέπει να το ελέγξουμε για την 24 παρακαλώ άρχεται πέρας 20 προς 25. Απορρίπτεται. Είναι καυτή η ψηφοφορία. Ε, η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε για 45 παρακαλώ πέρας 18 προς 24 απορρίπτεται η 46 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ άρχεται πέρας 25 προς 20 ψήφοι, εγκρίνεται η 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία φυσικά. Α, είναι μόνο γνωμοδότης, καλά. Απλή ψηφοφορία τότε. 40 προς 5 αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Βίρκουναν. Τώρα η γνωμοδότηση για το πρωτόκολλο του Παρισιού. Συμβαστική ένα είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Τροπολογία 2 παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Με 19 προς 25 απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Έλεγχος, δεν κατάφερα να, να το πω με σιγουριά, παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. 66 προς 9. Ε, πολύ δεν σήκωσαν το χέρι. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά. Από εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά Αποχέ και πάλι πρέπει να κάνουμε την επαλήθευση για τροπολογία 5. Άρχεται, πέρας. 30 προς 15. Συμβαστική 3, υπέρ. Κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Η τροπολογία 24, υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίψεται. Η συμβαστική 4, υπέρ. Κατά εσείς εγκρίνεται. Συμβαστική 5 είπε, κατά, εσείς εγκρίνεται. 31 είπε, κατά, εσείς απορρίπτεται. Συμβαστική 6 είπε, κατά, εσείς εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση για το 41 παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. 19 προς 22. Απορρίπτεται. Όχι 19 προς 23 τέλος πάντων. Συμβατική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 αποσύρεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Κλείνω ηλεκτρονικό την ψηφοφορία. 40 προς 3, δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κάνουμε μια σύντομη διακοπή μέχρι να έρθει ο Υπουργός γιατί ήμασταν πολύ γρήγοροι σήμερα. I think we can start. Πρόεδρος, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στα γερμανικά. Το επόμενο σημείο στη η για διάταξη και θέλω να χαιρετήσω τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Φρασού Μπάς, ο οποίος είναι αρμόδιος για το ε, μεταφορικό πακέτο. Θα μας εξηγήσει ποιες είναι οι προθέσεις του το επόμενο εξάμεινο για κάτι διάρκεια της Προεδρίας. Του κύριε Μπάους, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μίκαλ, με μεγάλη μου χαρά ήρθα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί ως Προεδρεύον του Συμβουλίου θα έχουμε μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της συναπόφασης αλλά επίσης και γιατί και ο ίδιος επί 24 χρόνια διετέλεσα βουλευτή πριν ε, αναλάβω τα πολιτικά καθήκοντα, οπότε ξέρω τα του κοινοβουλευτικού βίου. Οπότε, ξέρω καλά ότι θα πρέπει κανεί να σέβεται το κοινοβούλιο και οπότε έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή με το κοινοβούλιο ε, γιατί πολλές φορές αυτό δεν είναι στην πολιτική αυτονόητο αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό οπότε μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σα σήμερα για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας. Μία προκτευτική παρατήρηση. Δεν λέω κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να αναδουλέψουμε για πέντε μήνες γιατί βγάζουμε τον Αύγουστο ε, οπότε εκεί τα πράγματα έχουν αργούς ρυθμούς ούτε επίσης θα τώρα έχω τα εξή 50 σημεία ως προτεραιότητε και στο τέλος της ε, Προεδρία να ξαναέρθω εδώ και να σας πω ε, τι να κάνουμε. Ε, είχαμε 50 θέματα και τελικά δεν πετύχαμε τίποτα πόδι γι' αυτό θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία σήμερα είναι τα πιο σημαντικά εκείνα τα οποία έχουν οριμάσει για να προωθηθούν σε μέσα επόμενους και πρώτα πρώτα έχουμε το τέταρτο πακέτο για του συνδρόμους. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την Λετωνική Προεδρία και οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το εξαίρετο έργο το οποίο ε, επετέλεσαν κατά και κατά το τέλος της Προεδρίας τόσο ώστε από τεχνικής πλευράς να βάλουν τις τελευταίες πινελιές οπότε και εμείς τώρα θα επικεντρώσουμε τις προσοχή μας στα πολιτικά ζητήματα δηλαδή στα της ε, διακυβέρνησης και και στο PSO. Οπότε θα πρέπει να πετύχουμε κάποια συνένεση στους αμέσους επόμενους μήνες. Ίσως θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε αναρωτηθεί ποιος είναι ο στόχος ναι, για το πακέτο αυτό. Να έχουμε περισσότερου ισοδρόμου, καλύτερη ποιότητα, καλύτερη αποδοτικότητα στην Ευρώπη στον αφορά Να, ποιο είναι ο στόχο μα. Οπότε νομίζω ότι τώρα, του επόμενου μήνε, θα πρέπει να ε, εργαστούμε με αυτό το πνεύμα έχοντας υπόψη αυτό τον στόχο να αναζητήσουμε μια συνένεση και έτσι να ε, λάβουμε υπόψη τις ιδιοτυπίες του κάθε κράτους μέλους και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική επιτυχία θα καταλήξει σε κάποια συμφωνία τον ε, Οκτώβριο, 8 Δεκάτου το Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο. Στόχος να το λίγο αργότερο. Οπότε αυτό το συνολικό πακέτο είναι ένα θέμα προτεραιότητας. Οπότε και η Προεδρία με αυτό θα ασχοληθεί στους επόμενους μήνες. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η αεροπλοεία. Δεν χρειάζεται να εξηγώ σε ευρωβουλευτές πού έγκυται οι δυσκολίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Τα ξέρετε καλύτερα και από μένα και γνωρίζετε ότι δεν είναι μόνο θέμα υπουργών μεταφορών, είναι θέμα πολιτικής γενικότερο και τη σημερινή μέρα είναι πολύ δύσκολο το να προωθεί ο φάκελος αυτό το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, Είμαστε πραγματικά πεπισμένοι ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα. Και υπάρχει και ένα σημείο επί το οποίο το Κοινοβούλιο το έχει πάει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Είναι το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών και θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έχει γίνει και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε, θα έλεγα άτυπα, για όλα τα επιμέρους θέματα της ε, αεροπλοείας ή των αερομεταφορών όλα αυτά που θα απασχολήσουν την Προεδρία μα Με τα πολιτικά ζητήματα και ζητήματα τα οποία δεν είναι δική μου αρμοδιότητα γιατί είμαι υπουργό μεταφορών. Όμω, σα διαβεβαιώ ότι στον τριμερή διάλογο ε, δουλεύουμε ομαδικά. Τα πήγαμε πολύ καλά με την Λετωνική Προεδρία αλλά και με την Ολλανδική Προεδρία την Οπότε, ήδη έχουν γίνει σημαντικέ συζητήσει με του Ολλανδού συναδέλφου. Σα διαβεβαιώνω ότι έχουν κάθε πρόθεση να εμπιστατεύσουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσουμε. Ας πούμε βέβαια, να κάνουμε τον Ιανουάριο ένα τύπο συμβούλιο όσον αφορά ε, σε αεροπορικές μεταφορές. Το είναι πολύ σημαντικό. Ένα τρίτο θέμα το οποίο έχει σχέση με την διάσκεψη COP21. Είναι τα θέματα του περιβάλλοντος. Εκείνα τα οποία έχουν σχέση με τις μεταφορές. Και πρώτα να δούμε αυτού του τον καταστροφικό υπολογισμό, απολογισμό που ισχύει σήμερα, δηλαδή το ότι οι μεταφορέ είναι ο μόνος κλάδος σήμερα όπου οι εκπομπές του διοξιδίου δεν έχουν μειωθεί, έχουν αυξηθεί 20%. Αν αναχθούμε στην περίοδο μέχρι το 90. Οπότε έχουμε τη διάσκεψη αυτή των Παρισίων. Και οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα καταβάλουν κάποιε προσπάθειε για τι μεταφορέ και άρα θα μα απασχολήσει και αυτό. Άλλο σημείο πολύ σημαντικό θα θέλαμε και επ' αυτού να προσπαθήσουμε είναι η Λευκή βίβλο για τι μεταφορέ. Το κοινοβούλιο με τον κύριο Φαντεκάμ που βρίσκεται εδώ ενώπιόν μου Επιτέλεσε πολύ αξιόλογο έργο. Μου είπατε ότι μόλι έγκρινατε την έκθεση όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση τη Λευκή Βίβλου. Οπότε θα ήθελα να σα συγχαρώ για το έργο σα και για την έγκριση τη έκθεση. Οπότε η Προεδρία μας πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, αν όχι ε, μία συγκεκριμένη έκθεση, αλλά τουλάχιστον κατά τις συνεδριάσεις του, στις 8 ε, 10 του Λουξεμβούργου ιδίως να συζητήσει το ζήτημα αυτό της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης της Λευκής Βίβλου. Και ίσως κατόπιν της συζητήσεως και σφαντικά δεν προβούμε σε κάποια κοινή δήλωση, κοινή ανακοίνωση. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, άλλο επενδύσεις για τις υποδομές. Έχουμε βέβαια ευτυχώ το σχέδιο Γιούγκερ. Έχουμε τα ισχυρά κοινότητα του Κοινοβουλίου. Οπότε και εδώ θα καταβάλουμε προσπάθειες. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές επενδύσεις στις ε, υποδομές των μεταφορών. Είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα οικονομικού οράματος για τις μεταφορές. Αλλά να δούμε πώς θα καλυφθεί το ζήτημα αυτό στις εργασίες μας. Κάτι άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το καινούργιο. Θέλουμε να συμβιαλέσουμε στις 7 Δεκάτου στο Λουξεμβούργο ένα άτυπο συμβούλιο. Μία μέρα πριν την επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 8. Κάτι να δούμε για την κινητικότητα στις πόλεις και πιο συγκεκριμένα να δούμε τι γίνεται με τη χρήση του ποδηλάτου. Του ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς στην κοινωνία μας. Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι έχετε μια τροπολογία που αποσκοπεί ακριβώ σε αυτό, όπω μου είπατε, στα πλαίσια του κειμένου για τη Λευκή Βίβλο. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Είμαι πεπισμένο. Πώ μέχρι σήμερα έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ την υπόθεση του ποδηλάτου ω μέσο μεταφορά. είναι θέμα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της κινητικότητας της ε, πόλης που ξέρουμε πόσα προβλήματα τις μαστίζουν. Οπότε παρακαλώ να παρακολουθήσετε τις εργασίες ε, και την πρόοδο των εργασιών τέλο πάντων σε αυτό το άτυπο συμβούλιο του Συμβουλίου. Έχουμε τον Γιάνν και άλλους ε, ποιοτικού αγορητές εκεί προσκαλέσει που είναι πρόκειται από την Κοπενχάγη, ε, τον κύριο Κόλμπεν επίσης ο οποίος ε, έχει δώσει μάχες για την πρόθεση της υπόθεσης ε, ποδήλατο στην Ευρώπη. Τώρα κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα και αυτό να το καλύψουμε τις συζητήσεις μας για Λευκή είναι η οδική ασφάλεια. Και σε εθνικό επίπεδο αυτό με έχει απασχολήσει. Άρα νομίζω ότι την υπόθεση της οδική ασφάλειας μπορούμε να την εντάξουμε στις πολιτικές μας και την κοινωνική πτυχή του θέματος και την περιβαλλοντική. Όλα αυτά θα καλυφθούν από την προβληματική για την Λευκή Βίβλο. Με ενδιαφέρει το θέμα. Άλλο. Θέλουμε να απασχολήσει σε κάποιο επίσημο ε, συμβούλιο τον Δεκέμβριο η κοινωνική πτυχή του θέματος των δικών μεταφορών. Δύσκολο θέμα, το γνωρίζω. Δεν θέλω να το συζητήσουμε σε σχέση με την καινούργια νομοθεσία που θα θεσπίσουμε στην Ευρώπη. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Άρα θα είναι ενδιαφέρον αυτό να συζητηθεί το Δεκέμβριο σε ένα συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ βασικό το ότι ήδη επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πακέτο μέτρων για τις οδικές μεταφορές για το 16. Τώρα όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς και αυτό θα μας απασχολήσει, θα το βλέπουμε θετικά γιατί η Λετωνική Προεδρία τα πήγε πάρα πολύ καλά με το φάκελο αυτό. Οπότε και ταχαίως γίνονται οι διοργανικές επαφές, οπότε και νομίζω ότι εύκολα θα μας προκύψει πάνω σε αυτό μια συμφωνία. Με το Κοινοβούλιο τώρα όσον αφορά τις καταθάλασσες μεταφόρες και κυρίως τις ε, υπηρεσίες των λιμένων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σας, να δούμε πότε θα ολοκληρώσετε την πρώτη ανάγνωση που ήρθανε μέσα Δεκεμβρίου. Οπότε και κατά την εντολή μας, κατά την, το εξάμεινό μας θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να έχουμε μια συνάντηση και τα κράτη-μέλη να αποφανθούν όσον αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο. Τώρα, για τον τουρισμό. Και αυτό είναι η αρμοδιότητά σας. Έχουμε την κυρία Κλάους, που είναι η υφυπουργός μου. Ε, εκείνη χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο και θα σας την στείλω. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα θεματολόγιο πολύ πλούσιο για τους επόμενους μήνες. Αυτά θα μας απασχολήσουν τους υπουργού μεταφορών στο Συμβουλίο. Οπότε και ελπίζω πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Και περιμένω πώς και πώ τις τείχων ερωτήσει αλλά και τι προτάσεις vielen Dank, Herr Minister Bausch. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάους. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και τώρα θα αρχίσει ο διάλογος με τους συντονιστές πρώτα, 2,5 λεπτά οι συντονιστές λόγω πίεσης χρόνου και ενάμιση για τους λοιπούς ομιλητές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έλευσή σας και την παρουσίασή σας. Ο Βιν Φαντεν Κάμπ είναι ο πρώτος ο οποίος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτού προχωρήσω περαιτέρω, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Υπουργό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την σαφήνεια το, της παρουσίασής σας. Εγώ έχω κάθε εμπιστοσύνη στις προεδρίες των μικρών χωρών. Το είδαμε αυτό και στη Λετωνική Προεδρία, πόσο καλά κάναν τη δουλειά τους και πιστεύω ότι και το Λουξεμβούργο θα μπορέσει να συνεχίσει σε αυτή την ίδια κατεύθυνση. Και έχω και άλλες ελπίδες τις οποίες τρέφω, γιατί μετά το Λουξεμβούργο θα αναλάβει τη σκητάλη η Ολλανδία, οι 100 Θα είναι πολύ θετικό αν οι Λουξεμβούργοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καυτά θέματα και να διευκολύνουν το έργο των κατοχωρητών μετά. Σίγουρα πρέπει να εστιάσετε στο τέταρτο συνδεδομικό πακέτο και τα θέματα της αεροπλοΐας. Για το τέταρτο σιδηροδομικό πακέτο, η πολιτική πτυχή αυτού του πακέτου αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα. Το τόνισα προηγουμένως. ότι η, η βέλτιστη λύση είναι ο αντίπαλος της της εφικτής λύσης. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει μια εφικτή λύση, γιατί δεν νομίζω θα μπορέσουν να περάσουν όλες οι ρήτρε του τέταρτου πακέτου εφέτος. Όλα αυτά εξαρτώνται και από τις ε, ανάγκες για τον τεχνικό πυλώνα, για τη διάσκεψη των Παρισίων. Ξέρω ότι έρχεστε από τους πράσινους κύριε Υπουργέ, <clears throat> αλλά προτού δαπανίσει κανείς τα χρήματα πρέπει να τα βρει πρώτα. Και το ΕΛΚ θέλει να δώσει την πρέπουσα προσοχή στο γεγονός ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήματα στον τομέα των μεταφορών. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώνουμε μονάχα για να πετύχουμε. Δύσκολο να πετύχουμε αυτήν την ισορροπία, αλλά ελπίζω ότι το έχετε υπόψη Και μετά για τη συνάντηση της 7ης Οκτωβρίου. Θα πάτε εσείς με το ποδήλατο και ο ίδιος ή απλώς κάνετε διαφήμιση για τα ποδήλατα. Φαίνεται ότι ο κύριος Κράμερ είναι ο μόνος πεπισμένος ποδηλάτης. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και από σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έρτου. Κύριε Υπουργέ, και από την πλευρά της Σοσιαλιστικής Ομάδος θέλω να σας καλωσορίσω στην συνεδρίασή μας ή στην Επιτροπή Μεταφορών. Εγώ Χαίρομαι ιδιαίτερα βέβαια που έχω απέναντί μου ένα πράσινο υπουργό και έρχεστε από ένα μεγάλο σημαντικό κόμμα στο Λουξεμβούργο, κάτι που μου δίνει περαιτέρω χαρά. Αναφερθήκατε σε σημαντικά θέματα από το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο μέχρι τα θέματα της αεροπλοείας. Είναι όλα αυτά σημαντικά θέματα. Σας, ελπίζω, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για τα ζητήματα αυτά, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ιδίως για το τέταρτο πακέτο ε, για τα συνοδευτικά θέματα είναι μια καυτή πατάτα, όπω είπε και ο κύριος Φαντενκάμπ. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για τα τεχνικά θέματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση, αλλά τα πολιτικά θέματα είναι κάπω πιο δύσκολα από ότι στο παρελθόν. Θα, δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί μια λύση, γιατί πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία αντιμετωπίζει και τι ιδιαιτερότητε των κρατών μελών. Δεν είναι αδύνατον αλλά δύσκολο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, τον αεροπορικό κλάδο, η προστασία των επιβατών είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και η δική μου ομάδα, και όχι μόνο η δική μου ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδιαφέρεται ώστε το πακέτο για, την, ε, για τον αεροπορικό κλάδο να μπορέσει μέχρι το τέλος του έτους να έρθει η ψήφιση και να περιλαμβάνει και να μια λύση σε διάφορα σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή μας φαίνονται προβληματικά όπως είναι παραδείγματος το pay to flying, το wet leasing, το leasing των αεροσκαφών μαζί με το, με το πλήρωμά του, τις εταιρείες γραμματοκιβωτίου κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία υπονομεύουν τις κοινωνικές συνθήκες στον τομέα του αεροπορικού κλάδου. Περιμένουμε λοιπόν από τη Λουξεμβουργική Προεδρία να κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες για μας ε, ως σοσιαλιστές θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε επίση το θέμα της, των μεταφορών ως συντελεστή για την οικονομική ανάπτυξη και εκεί δυστυχώς βλέπουμε ότι όπως και στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά κράτη-μέλη θεωρείται ότι είναι ένας δευτερεύον τομέας ο των μεταφορών. Αυτό είναι κρίμα και είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε ώστε να ενισχύσετε στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών τη σημασία της κινητικότητας και των μεταφορών και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συγκοινωνιών και στον κοινωνικό τομέα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλή τύχη. Ο Ρόμπερτ Ζήλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας από πλευράς των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Είμαι από τη Λετωνία, από μια μικρή και χωρίς μεγάλη εμπειρία χώρα. Αντίθετα, εσείς έχετε αναλάβει την Προεδρία πολλές φορές. Και έχουμε μεγάλη ε, εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας. Σε σχέση με το πρόγραμμά σας και το τέταρτο συνδρομικό πακέτο, θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. εφόσον φαίνεται ότι το έχετε αναδείξει σε προτεραιότητα. Ε, Τον Οκτώβρη ε, θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Μεταφορών στο Συμβούλιο και εκεί θα συζητηθούν πολιτικά ζητήματα και θεωρείτε λοιπόν ότι μπορείτε και στην πράξη κάτι να κάνετε στους τέσσερις μήνες που θα έχουν απομείνει εάν επέλθει πολιτική συμφωνία για τα τεχνικά μέτρα. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή γιατί χρειάζεται την πολιτική εντολή. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια σε σχέση με το τι θα συμβεί ε, στο Συμβούλιο Υπουργών του Οκτωβρίου. Εάν για τις πολιτικές ψυχές ε, καταλήξετε σε συμφωνία, θέλω να ελπίζω ότι θα καταλήξετε και σε μια τεχνική συμφωνία. Είναι λεπτό το ζήτημα και δίστατη και απόψε εδώ στην Επιτροπή μας σε σχέση με το πόσο αυστηρή πρέπει να είναι κάθε νομοθετική ρύθμιση Υπάρχει το θέμα του ελαχίστου μισθού. Δεν έχει, έχει μεγάλη διαφορά ελάχιστος μισθού στη Λετωνία και τη Βουλγαρία, παραδείγματο χάρη. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια ισορροπία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη θεωρία έχουμε μια εσωτερική αγορά όπου ισχύουν ομοιόμορφες ε, συνθήκες για την εργασία, στην πράξη όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ε, ως προς το σχέδιο Juncker για τις μεταφορές, γιατί ασχολήθηκε και με αυτό η Επιτροπή μας, διαπιστώνουμε ότι έχουν έχει υπάρξει δηλωμένη υποστήριξη για κάποια προγράμματα, και υπάρχει διαφορά από τα μέτρα που προξένει η δική μας Επιτροπή. Πώς το βλέπετε εσείς, ε, ποια μέτρα θα προωθήσατε. Σας ευχαριστούμε και Ζήνα Μάεθα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ ε, να σε ευχαριστήσω ε, προσωπώ τους φιλελεύθερους. Χαιρόμαστε εκ των προτέρων για την Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Όπως είπε ο συνάδελφος Τσίλε, είστε μια μικρή χώρα, όμως έχετε ευρύτατη εμπειρία δεν θυμάμαι καν πόσες φορές έχει αναλάβει την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Τέλο πάντων, έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε. Ε, είναι πολύ σημαντικό το συνδυναμικό πακέτο για την Ευρώπη και το ξέρετε, οπότε ε, θα ήταν σημαντικό την πρώτη τεχνική πτυχή να την υλοποιήσουμε, να τη συμφωνήσουμε για να την υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Διότι... Διότι διότι ε, αυτό το χρειαζόμαστε πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα τα καταφέρετε λοιπόν να εξασφαλίσετε ότι για το θέμα του βράχου του Γιβραλτάρ δεν πρέπει να έχουμε διαμάχες για θέματα κυριαρχίας, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις αεροπορικές συνδέσεις. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσετε να το κάνετε και να εξασφαλίσετε και τα δικαιώματα των, των επιβατών των αεροπορικών γραμμών. Σε σχέση με το Connecting Europe, εσείς ξέρετε ως Λουξεμβουργέζος για το σχέδιο ε, Juncker, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά χρήματα τα οποία έχουν φύγει από το τομέα των μεταφορών στο ΕΦΣΥ. Αυτό σημαίνει για μας όμως ότι θα πρέπει να τύχουν κάποιες υποστήριξεις στα σχέδια μεταφορών στο πακέτο Juncker. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχετε κάποιο βλέφαρο στα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσει να γίνει πράγματι, πραγματικότητα, να ενσωματωθούν και τα σχέδια ε, μεταφορών και επίσης ότι θα υπάρξουν αρκετές ενέργειες στο τομέα των εσωτερικών πλωτών οδών, ώστε να μπορέσουμε στο βαθμό του δυνατού να μεταφέρουμε κίνηση από τους δρόμους στις εσωτερικές υδάτινες οδούς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, για τα ποδήλατα. Εγώ σας ε, συγχαίρω απόλυτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια συνδιάσκεψη η οποία να είναι φιλική προς το περιβάλλον και για, την οδική, ε, για τα οδικά θέματα δεν είπατε τίποτα για το Uber αλλά θα περίμενα να πείτε κάτι. Ευχαριστώ η Μάγια Κίλενεν έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να... Ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για το σιδηροδρομικό πακέτο. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στον τομέα των μεταφορών αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση. Να εστιάσετε την προσοχή σας ε, κατά προτεραιότητα σε αυτό το πακέτο, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Είναι σημαντικό, όπως και το πρόγραμμα για τον Ευρωπαϊκό Ουρανό, για την ασφάλεια στη, στον τομέα των αερομεταφορών. Για όλα αυτά, σημαντικό ε, είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης. Όμως, ξαναλέω, επαναλαμβάνω πόσο σημαντικό είναι το σειροδρομικό πακέτο. Ελπίζουμε να υπάρξει και ισότιμη μεταχείριση για όλα τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των πολιτικών ζητημάτων. Σας ευχαριστώ ε, Είναι στο νοσοκομείο ο από τους Πρασίνους. Ε, ε, τελειώνουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση. Εσείς μίλησατε για το 20% μείωση των εκπομπών στις, ε, στις μεταφορές. 20% στη βιομηχανία έχει γίνει πραγματικότητα, αλλά στις πόλεις τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Όλες οι, 70% των εκπομπών που είναι αρνητικές για το κλίμα προέρχονται από τις αστικές μετακίνησεις. 90% των αυτοκινήτων στην Γερμανία, είπε ο Γερμανός Υπουργός, κινούνται για αποστάσεις μέχρι 6 χιλιόμετρα. Αυτό είναι πολύ καλό να το αντιμετωπίσει κανείς με το να ευνοήσει, το να πηγαίνει κανείς με το πόδι, με το ποδήλατο. Και βέβαια με το ποδήλατο πηγαίνει κανείς πολύ πιο γρήγορα από το ποδήλατο. Εγώ το βλέπω αυτό. Είναι η δική μου εμπειρία και όχι μόνο να κέρδιζε χρόνο, αλλά είναι πολύ καλό και για την υγεία. Μιλήσατε επίσης και για τον τουρισμό. Ο τουρισμός του ποδηλάτου όλο και περισσότερο δημιουργεί χρήματα. 44 δισεκατομμύρια ευρώ λέει όσο και τα κρουαζιερόπλια. Είναι πιο εύκολα βέβαια να πάρει κανείς χρήματα για τα κρουαζιερόπλια από ότι για την υποδομή των ποδηλάτων, αλλά είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό και στην άτυπη συνεδρίαση των ε, Βρυξελών. Εγώ χαίρομαι που θα μπορέσω να σας συναντήσω εκεί. Μιλήσατε επίση και για την εσωτερική, σειρά την οδού. Εμείς φυσικά υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο ως ε, πράσινη, αλλά θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπέ και υπάρχει και το θέμα της ε, διέλευσης από τα από τους υδατοφράκτες που περνούν τα πλοία. Και έχουμε τώρα αυτούς που έρχονται με διάφορα σχέδια με τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αλλά εκεί είναι το σημαντικό να δούμε που πρέπει να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Και επίσης για την διαμεθοριακή ε, μεταφορά είδα ότι υπάρχει μια συμφωνία Λορένης με, το, με τη Δυνανία Παλατινάτο έχουν κάνει μια συμφωνία ώστε να υπάρξει μια σύνδεση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το Λουξεμβούργο. Αυτό θα είναι πολύ καλό να έχουμε ένα σχέδιο τριών χωρών. Αυτό είναι πολύ καλό θετικό παράδειγμα και για το μέλλον. Ποιος ακολουθεί? Jetzt kommt äh, David Maria Sassoli. Sassoli. Grazie. Ευχαριστώ. Να μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα Υπουργέ. Ευχαριστούμε για τα όσα μας εξηγήσατε. Γιατί διευκρινίσατε το ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Εγώ είμαι συγγητής για την έκθεση του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου. Οπότε θα παρακολουθήσω από κοντά το έργο σας. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται την ε, ενθάρρυνση, οπότε και οι δικέ σα ε, ενέργειε θα είναι κάτι το οποίο θα μα απασχολήσουν. Θα, μεγάλη προσοχή θα ε, βλέπουμε τι κάνετε και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα φτάσουμε τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο Μεταφορών έτοιμοι για να δώσουμε μια όθηση στην υπόθεση τέταρτο πακέτο. Και έτσι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή που είναι τόσο σημαντική. Για πες τον παρακαλώ για σας. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο ενδεχόμενο συμβασμό στο Συμβούλιο, γιατί έχουμε εδώ πέρα του δύο φακέλου που αφορούν το τέταρτο πακέτο. Επίση και για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό είμαι εισηγητή για την διακυβέρνησή του και ξέρουμε ότι έχει επιφέρει την εμπλογή το Συμβούλιο γιατί υπάρχει αυτή η διχογνωμία για το Γιβραλτάρ, οπότε και αυτό το πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε είναι σε γενοτικό επίπεδο να προχωρήσουμε για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα των αερομεταφορών, το οποίο όπως ξέρετε ο ανταγωνισμός μας πιέζει και συγκεκριμένα από τα Εμμυράτα, από τις χώρες του κόλπου. Οπότε για πες μας τι προτείνετε να κάνετε σχετικά. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κριστίνα Βονταλόν. Merci, merci, monsieur le Ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Χαίρομαι που στο πρόγραμμα εργασίας σας διαβάζω πως η κοινωνική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών συνιστά σας προτεραιότητα. Χωρίς ισχυρή πολιτική δέσμευση δεν θα προχωρήσουν τα πράγματα, κυρίως στο τομέα των μεταφορών όπου βλέπουμε ε, όλη την ουσία των προβλημάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Λουξεμβούργο έχει καταδείξει τη δέσμευσή του στα πλαίσια μια κοινή δήλωση με άλλα κράτη-μέλη στι 5 Ιουνίου του 2014 για την καλύτερη εφαρμογή τη υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να ενθαρρύνει του κοινωνικού εταίρου να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για να καταπολεμήσουν ναι, τι ε, συνθήκε σε γραμματοκιβώτια και για να προωθήσουν ε, θεμητού όρου ανταγωνισμού. Ελπίζουμε λοιπόν να αναλάβετε και ηγετικό ρόλο για να ανταπεξέλθετε σε αυτές τις προκλήσεις. Φυσικά θέλω και εγώ να μιλήσω για την πολιτική πτυχή του σιδηροδρομικού πακέτου. Θα το έχετε ήδη καταλάβει ότι και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό και από ό,τι καταλάβαμε στην για σα προτεραιότητα σε αυτό το φάκελο ε, και την έκθεση των του Ιωνίου βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει για τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα. Ελπίζουμε ε, με την Προεδρία σα να σημειωθεί πρόοδο, ούτω ώστε ε, να μην θεωρήσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε για να είναι αποτελεσματική δρόμη να υπάρχει μεγαλύτερο άνοιγμα, να αφήσουμε στι αρμόδιε αρχέ την αρμοδιότητα για να οργανώσουν τι δημόσιε υπηρεσίε για να εξασφαλίσουμε την εδαφική συνοχή είναι απαραίτητο να μην οδηγηθούμε σε κατάργηση λιγότερο μεν αποτελεσματικών ε, διαδρομών, αλλά που είναι απαραίτητε για τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρε διατάξει για τα εξτάμενα κοινωνικά πρότυπα για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταφορών των εργαζομένων, απόσπαση των εργαζομένων ανάμεσα σε εταιρείε. Ευχαριστούμε, Μάρκο Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις προτεραιότητες που μας αναφέρατε. Ακούσατε από πολλούς άλλους πόσο σημαντικό είναι το πακέτο για τα σιδηροδρομικά θέματα. Τι θα γίνει όμως θα ήθελα να ρωτήσω αν δεν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία. Τι θα κάνετε με την δική σας θητεία. Δεύτερον, το θέμα της ε, ποδηλασίας. Οι κάτω είναι ο παράδεισος των ποδηλάτων και το Μούνστερ στη Γερμανία είναι επίσης αντίστοιχο, η αντίστοιχη περιοχή στην ε, Γερμανία. Αυτό οδήγησε σε κάποια αλλαγή νοοτροπίας από την πόλη μας, την περιοχή μας. Αν βλέπω λοιπόν την έννοια αυτού του διαδρόμου από την Ολλανδία ως την ε, ε, Βαρσοβία είναι σημαντικό να υπάρξει μια διεθνής διάσταση σε στο άνοιγμα δρόμων. Μήπως λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε θέμα εθνικού επίπεδου. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές και τη μεταλαμπάδευση τους. Γιατί πάνε τόσο καλά τα πράγματα στις κάτω χώρες. Αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι με υποχρεωτικούς κανόνες και με πιέσεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και τότε με τους ε, πεζούς. Είναι υπερβολικές όλες αυτές οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Καλά είναι αυτά που λέτε για το, την εναέρια κυκλοφορία και τους ποδηλάτες, αλλά ίσως ανεδαφικά. Λουκατσέφσκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η κοινωνική διάσταση των οδικών μεταφορών. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα. Στην διάσκεψη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, κοινωνικό θεματολόγιο για τις μεταφορές, μας μιλήσατε για αυτή την ε, σύγχρονη δουλεία των ε, οδηγών φορτηγών και συμφωνώ μαζί σας, ε, είμαι υπέρ της ε, καταπολέμησης όλων των καταχρήσεων σε αυτό το τομέα στα πλαίσια ε, όμως ε, τη ενίας αγοράς ε, υπάρχουν πολύ διαφορετικές αμοιβέ, ε, πολύ διαφορετική μισθή και δεν είναι δυνατόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει πλήρη εναρμόνιση. Δεν, δεν έχει νόημα να το επιδιώξουμε. Μιλώντας για, για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο μας είπατε ότι ένα από τους στόχους αυτού του πακέτου είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του των σιδηροδρόμων, λαμβάνοντας υπόψη όμως τι ιδιαιτερότητες ε, κάθε χώρας. Ελπίζω λοιπόν ότι και στα πλαίσια του, ε, των οδικών μεταφορών, παρά τις καταχρήσεις που υπάρχουν, θα λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όντως στην Πολωνία, στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία θα ήθελαν να έχουν ένα, μια αντίστοιχη αμοιβή όπως στο Λουξεμβούργο παραδείγματο. χάρη. Δυστυχώ προς το παρόν δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Η Φώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν οι θαλάσσιες μεταφορές. <clears throat> Νομίζω <clears throat> ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για τα καθαρά καύσιμα και τα καθαρά νερά. Έχουμε τώρα και το τομέα των κρουαζιεροπλοίων που έχουν να αντιμετωπίσουν στους εθνικούς κανόνες στα λιμάνια και το έχω θέσει το θέμα αυτό και στην Κομισιόν. Θα ήθελα η Προεδρία σας να βοηθήσει να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Για το πακέτο αεροπορικών συγκοινωνιών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα περάσουμε σε μια συζήτηση με, το, με τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και εγώ είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό και εδώ θέλω να θέσω μονάχα αυτή την παρατήρηση. Όλοι νιώθουμε μια ματέωση για τα θέματα της ε, ε αεροπορίας. Εγώ ήμουν η πρώτη εισηγήτρια για τους ενιαίους εθέρες. Η Μεγάλη Βρετανία ήθελε να προωθήσει το θέμα αυτό αλλά τελικά ό,τι και να γίνει το Γιβραλτάρ είναι ανεξάρτητο κράτος είναι έξω από την ενιαία αγορά, δεν μπορεί αυτό να τεθεί σε διαπραγμάτευση. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικός, υπάρχουν πολλά απλώς λόγια που λέγονται σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να φτάσουν και να κάνουν ε, συγκοινωνίες στην Ευρώπη το κοινωνικό dumping, αυτό που λένε πάρα πολύ, είναι μια, ένα πρόσχημα για προστατευτισμό. Εγώ έρχομαι από ένα νησί όπου ενδιαφερόμαστε για μια ανταγωνιστική αγορά. Ευχαριστώ λοιπόν. Ο Τζος Μπαχ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Φράνς. Θέλω να σας συγχαρώ για το φιλόδοξο πρόγραμμά σας και σας και την ομάδα σας έχετε αναφέρει τις προτεραιότητές σας και για το τέταρτο πακέτο για τα σιδηροδρομικά είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε να καταλήξετε σε μια λύση η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, θα ικανοποιήσει τους πελάτες και τις επιχειρήσεις. Έχετε επίσης αναφερθεί στις κοινωνικές πτυχές των οδικών μεταφορών και τονίσατε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή των ελέγχων και των ενδεχομένων, ενδεχομένους κυρώσεων. Σήμερα στην Λευκή Βίβλο, στην ψηφοφορία μας, έχουμε ζητήσει να υπάρχει ένας φορέας για την οδική μεταφορά, η οποία περιλαμβάνει ε, και αυτές τις δυνατότητες και τα συνδικάτα και οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απάντηση στο γράμμα μας και λέτε ότι εσείς προσπαθείτε να δείτε πώς μπορείτε να προωθήσετε και τα θέματα ουσίας Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες και υπήρχε και ένα ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Είσαστε φυσικά και υπουργό για βιώσιμη ανάπτυξη εσείς. Γι' αυτό σας ρωτώ ποια είναι η άποψή σας για τα θέματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας και πώς λοιπόν θα κινηθείτε σε σχέση με την οδηγία για τη μείωση των εκπομπών από τα οχήματα και την πρόθεση των προτύπων Euro 5 και 6. Και αν έχετε μια ανοχή 10 δευτερολεπτών, το 2013 είχατε αναφερθεί και στα θέματα βαρέων οχημάτων και ασφάλειας στους δρόμους. Η Κομισιόν παραμένει ακόμα την ε, επιζήτηση αυτού του στόχου για να μειωθούν τα θύματα στους ε, δρόμους και δεν μιλάμε μονάχα ε, για, τα, για τους νεκρούς αλλά και για τους βαριά τραυματισμένους. Μπορείτε λοιπόν να πιέσετε την Κομισιό να προωθήσει και πάλι αυτό το θέμα. Είμαι κάπως πιο ανεκτικός για τους Λουξεμβουργέους, αλλά τα δέκα δευτερόλεπτα τα περάσατε παρασάγκα. Σήμερα είμαι όμως γενναιόδωρος, λέει ο Πρόεδρος και έτσι μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ. Α, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ε, συγχαρώ. κυρία Μπαραντίκα είναι αυτή. Τέλος, ευχαριστώ λοιπόν και για τα ε, σχέδιά σας για το επόμενο εξάμεινο. Θέλω να επικεντρωθώ στα σημεία τα οποία αναφέρατε ως προτεραιότητες της Λουξεμβουργικής Προεδρίας θα ήθελα να σας ζητήσω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να μπορέσετε να προωθήσετε συνεκτικά όλα αυτά τα θέματα. Γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρετε είναι αλληλένδετα. Αν εμείς δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε οδηγίες και κανονισμούς που έχουμε ήδη εγκρίνει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. <coughs> ποτέ δεν θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό χάρτη διατροπικών μεταφορών όπου όλες οι μορφές μεταφορών έχουν μια σύνδεση μεταξύ τους και μπορεί ο επιβάτης με ένα μοναδικό εισιτήριο να κινείται από τη μια άκρη στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να εξασφαλίσετε τη συνεκτικότητα των νομοθετημάτων. Αν μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις υποδομές, και να τις κατασκευάσουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του, των εθνικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να δει ο πολίτης ότι η Ευρώπη είναι χρήσιμη. Είναι ένα μήνυμα το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό. Τούτου λεχθέντος επίσης θα πρέπει να μειώσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος γιατί συνέχεια μιλάμε για εκπομπές, τι μπορούμε να κάνουμε στις εκπομπές αλλά υπάρχει μια έλλειψη συνέπειας και συνοχή στην πολιτική μας που οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών. Για να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι σας συγχαίρω που θέτετε ως προτεραιότητα το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο μέσα στα πλαίσια των πολιτικών μας θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε μια κοινή στάση για τα σιδηροδρομικά θέματα αλλά κυρίως θα πρέπει να ξεπεράσουμε και τις δυσκολίες στον πολιτικό πυλώνα για το σιδηροδρομικό πακέτο. Χωρίς αυτά λοιπόν δεν θα έχουμε συντεκτική πολιτική και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς αναφερθήκατε ότι θέλετε μια συμφωνία και εμείς θέλουμε μια συμφωνία. Μιλήσατε όμως για την ανάγκη να καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό παρακαλώ και μέχρι πότε μπορεί κανείς να φτάσει με αυτή τη λογική σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο Τούρμες ως προσκεκλημένο σήμερα. Ήρθα εδώ. Γιατί είναι ο υπουργό μου εδώ, λέει ο κύριος Τούρμες. Τρία ερωτήματα για την ποδηλατοπρωτοβουλία που είναι πολύ σημαντική για μένα. Στον τομέα της ενέργειας έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο ε, μέτρων για τις πόλεις. Έχουμε το σύμφωνο των δημάρχων οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για την προστασία του κλίματος. Το θέμα είναι για τις αστικές μεταφορές που είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα και για την πρωτοβουλία των ποδηλάτων και επέκεινα αυτής είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κινητικότητας στις πόλεις. Για το σιδηροδρομικό πακέτο. Εδώ δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ιδεολογικά. Η φιλελευθερωποίηση δεν είναι αυτός σκοπός. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα στις διαμεθοριακές ε, συγκοινωνίες. Αυτό σημαίνει πρέπει να αποφύγουμε και το κοινωνικό dumping. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσετε να βρείτε μια συμφωνία η οποία εγγυάται και για την ποιότητα και είναι κατά του κοινωνικού dumping. Αν σκεφτείτε το, τη διαδρομή ε, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Μιλάνο. Παλιά υπήρχαν δύο νυχτερινά τρένα και οχτώ ημερήσιες συνδέσεις πριν από δεκα χρόνια. Τώρα έχουν μείνει μόνο δύο. Με την ε, ατελή αυτή φιλελευθερωποίηση ψόφισαν τα τρένα. Δεν έχουν μείνει λοιπόν αρκετέ συνδρομικέ συνδέσει στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια νέα όθηση. Και το τελευταίο ερώτημα. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο σοσιαλιστή συνάδελφο το κοινωνικό dumping στα φορτηγά, στις μεταφορές με φορτηγά. Είναι απαραίτητο αυτό το οποίο έγινε στην ε, Γερμανία να υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός. Και τώρα τους ε, πάει στα δικαστήρια η Κομισιόν. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά στην Προεδρία σας. Η Μαρία Γραπίνη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Ε, πρόεδρε, για την ε, συνάντηση που οργανώσατε με τον, ε, πρόεδρο, με τον, συγγνώμη, από τον Υπουργό από το Λουξεμβούργο, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Και να περάσω κατευθείαν στην ουσία του ζητήματος, δηλαδή την ε, χρηματοδότηση δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε τα εμπόδια που υπάρχουν αποτελεσματικά και άρα δεν θα έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε προγράμματα αναβάθμισης των υποδομών και άρα την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ε, χρειάζεται ένα επαρκές δίκτυο υποδομών, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα μέτρα που προτείνονται μέσα στο σιδηροδρομικό πακέτο. Δυστυχώς δεν ε, λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικές προτεραιότητες και στην πράξη δεν νομίζω να έχουμε ε, τα ευκαιρία αποτελέσματα. Όπως είπε ο συνάδελφος, αναρωτιέμαι και εγώ με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Επιτροπή να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν ε, στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη. Εντάξει, ε, υπάρχει ένα ελάχιστο μισθό στη Γερμανία και στη Ρουμανία έχουμε πρόβλημα διότι υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται σε αντίστοιχη εταιρεία στη Ρουμανία και όταν μεταφέρονται στην Ρουμανία δεν έχουν πλέον τον ελάχιστο μισθό. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Και πώς μπορούμε να μην κάνουμε επενδύσεις στις υποδομές και να περιμένουμε ότι θα έχουμε ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε, Κόσμος Λουτόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Μα είπατε το θεματολόγιο τη προτεραιότητα και αναφέρατε και τι αερομεταφορέ μεταξύ αυτών. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούμε με προσοχή το τι κάνουν ε, οι άλλε χώρε και θέλουμε επίση να προσέχουμε μπα και επιδοτούν, παραεπιδοτούν τι αεροπορικέ εταιρείε. Γιατί αν θέλουν να το πράξουν αυτό θα πρέπει να το κάνουν σύμφωνα με κάποιου κανόνε και να υποστούν τις σχετικές συνέπειες. Ας πούμε αυτό ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις, αυτό ισχύει και για την πολωνική κυβέρνηση και την πολωνική ε, αεροπορική εταιρεία. Εάν υποσυντρέχει μια τέτοια περίπτωση, τότε θα πρέπει η εν λόγω εταιρεία να ε, λάβει κάποια μέτρα, θα πρέπει να περικόψει κάποια ε, δρομολόγια ακόμα και να επικερδεί. Οπότε θα πρέπει το ίδιο να ισχύσει και για τι αεροπορικέ εταιρείε και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, λειτουργούν με τα δεκανίκια της κρατικής ενίσχυσης. Έχουμε ας πούμε αυτό να ισχύει για τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι πρεσβεύει η, η Προεδρία αν προτίθεστε να λάβετε κάποια τέτοια μέτρα εις βάρος ευρωπαϊκών εταιριών. Ο και άλλοι τρεις και μετά τελειώνουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας Υπουργέ. Εγώ εκπροσωπώ την ε, πολιτική ομάδα Ευρώπη των Έθνων και ελευθερία Είπατε ότι δεν θέλετε να βάλετε πάρα πολλές ε, προτεραιότητες. Εγώ όμως μέτρησα 11. Πολλές δεν είναι για 5 μήνες. Τέλος πάντων, επισύρω την προσοχή σας σε τρία σημεία που θεωρώ σημαντικά. Εγώ εργαζόμουν επί 30 ετία σε μια αεροπορική εταιρεία τη Γαλλία, οπότε αυτό το θέμα των αερομεταφορών με ενδιαφέρει και με καίει. Οπότε θα ήθελα να σα πω ότι εδώ στην Επιτροπή μα αποδίδουμε σημασία στα δικαιώματα των, ε, ε, των ε, επιβατών, αλλά και στην ασφάλεια κυρίω των επιβατών. Οπότε, πέστε πάνω σε αυτό Πού βρίσκονται οι σχετικέ διαπραγματεύσει για τι αεροπορικέ μεταφορέ. Δεύτερο σημείο, έχουμε θίξει πάρα πολλέ φορέ τι γεωνικέ πτυχέ και γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε θέμα τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι έντονο φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά κυρίω του απεσπασμένου εργαζομένου. Επίση, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που μα αναφέρατε σχετικά με το ποδήλατο, το οποίο θα έπρεπε να είναι το μέσο μεταφορά στο πιο βασικό στην κοινωνία μας. Προσέξτε όμως κύριε Υπουργέ, διότι στην Γαλλία όπου και εξελέγεν, διαπιστώσαμε ότι αυτή η πολιτική που κατηγορεί το το ταχύ για την ε, μόλυνση και μπλοκάρει τα κέντρα των ε, ε πόλεων τελικά παραλύει την τοπική οικονομία και τα μικρομάγαζα. Οπότε αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι ανηλικρινέ, είναι φαρισαϊκό γιατί έχουμε τι δημόσιε μεταφορέ, βέβαια έχουμε και το ποδήλατο. Όμω όσον αφορά τι δημόσιε μεταφορέ στην ε, Γαλλία δεν έχουμε ρυθμίσει ούτε το θέμα τη έφτακτη λειτουργία ούτε τη ασφάλεια για τι δημόσιε μεταφορέ. Οπότε τότε να μπορούν οι οδηγοί των γεωταχή κάπου να παρκάρουν το αυτοκίνητό του και να τι χρησιμοποιήσουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Μπάους. Μιλήσατε για την, για την οδική ασφάλεια. Και εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε υποστηρίξει το στόχο της μείωσης των θανάτων στο δρόμο, αλλά επίσης όπως είπατε και πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός των βαριά τραυματισμένων. Εγώ όμως ε, αναρωτιέμαι αν η Κομισιόν θέλει να υποστηρίξει κάτι τέτοιο και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Αν υποστηρίζετε εμά ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσατε επίσης και για τα δικαιώματα των επιβατών στην αεροπορία αλλά και στις θαλάσσι, θαλάσσιες μεταφορές και τις οδικές μεταφορές. Εγώ είχα τονίσει πριν από μέρες ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι οι Ευρωπαίοι να μπορούν με ένα εισιτήριο να κινούνται σε όλη την Ευρώπη, αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα εισιτηρίων για διατροπικές μεταφορές. Θα μας υποστηρίξετε λοιπόν για αυτήν την ενιαία μεταφορά, ενιαίο εισιτήριο για μεταφορές στην Ευρώπη. Μαριάν Μαρινέσκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία που αναλάβατε να έρθετε εδώ για να συζητήσουμε τα θέματα του πακέτου μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικό. Έχω να σας πω ότι είστε κατοχυρωμένος από την συνθήκη. Όμως θα έπρεπε ήδη εδώ και πολύ χρόνο να έχει αρχίσει το Συμβούλιο τους τριμμένους διαλόγους. Προβλέπεται ειδική πλειοψηφία και όχι η ομοφωνία και προς το παρόν μόνο ένα κράτος μέλος έχει λάβει θέση. Άρα, προσέξτε τη λέει συνθήκη. Επίσης, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε όσον αφορά τον προπολογισμό Σίγουρα εμεί θα ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια τόσο ώστε να καλύψουμε όλα αυτά τα οποία αφιερέθησαν το Horizon 2020 και από το Connecting Europe Facility. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια κονδύλια το κοινοβούλιο τόσο ώστε να υπάρχουν εγγύσεις από το ΕΦΣΙ. Ό,τι προβλέπουμε αυτό για το ΣΕΦ. Οπότε παρακαλούμε βοηθήστε μας κατά αυτό. Ακόμα και αν πρόκειται να γίνει αυτό ει βάρο κάποιων χρηματοοικονομικών μέσων. Ο επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Λέει κύριε Ντέλη. Και εγώ όπως οι συνάδελφοι να σα ευχηθώ καλή επιτυχία. Μιλήσατε στην εισηγησή σα για τα κοινωνικά θέματα. Θέματα καυτά δηλαδή. Ε, επίσης, μα είπατε ότι δεν έχετε ε, πρόθεση να ε, θεσπίσετε καινούργια νομοθετήματα, αλλά θέλετε απλώς να εφαρμόσετε τα υπάρχοντα καλύτερα. Οπότε για πέστε μου περισσότερες λεπτομέρειες. Τι μηχανισμός θα μετέλθετε, τι θα κάνετε με κάποιες τυχόν πρωτοβουλίες τόσο ώστε να εφαρμόσετε την ισχύουσα νομοθεσία. θα κάνει η Προεδρία. Τώρα όσον αφορά το συνδρομικό πακέτο, εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για αυτήν την τέταρτη δεσμή με τον οπότε και εγώ θα συμφωνήσω με τους δύο προλεξάντες συναδέλφους που είπαν ότι θα ήταν καλή ιδέα εάν μπορούσε το Συμβούλιο να συμπήξει συμβιβασμό. Οπότε και θα ήθελα πάρα πολύ να μου εξηγήσετε τι περιθώρια συμβασμού υπάρχουν πέρα από τα όσα καταφέρει η Λιτωνική Προεδρία. Μπορείτε και εσείς να επισημάνετε κάποια σημεία που μπορούμε τελικά να τα βρούμε. Αυτά ήταν λοιπόν τα ερωτήματα. Και τώρα για 15 λεπτά έχετε δυνατότητα να δώσετε απάντηση σε όλα αυτά. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο. Νομίζω ότι ήταν παρεμβάσεις χρήσιμες. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί εξέφρασαν τι διάφορες ευαισθησίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερα κατά την παρουσίασή μου. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω προσωπικά σε κάθε ένα από τους ομιλητές. Θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω τα θέματα εκτός από μία ή δύο ειδικέ ε, παρεμβάσεις που δεν μπορώ να τις ε, αντιμετωπίσω ομαδοποιημένα. Για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Ο κ. Πίπερ μου είπε, μα τι θα κάνετε αν δεν υπάρξει συμφωνία στο, 8 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρξει συνένεση σε σχέση με το σιδηροδρομικό πακέτο στον πολιτικό πυλώνα. Ναι, είμαι ειλικρινής. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μου. Η δική μου προσέγγιση είναι θετική. Εγώ θέλω να προχωρήσω προς τα εμπρός και όχι να θέσω αμφιβολίες και ερωτηματικά στον εαυτό μου τι θα γίνει αν αποτύχω. Γιατί πιστεύω θα πετύχω. Δεν θέτω αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εργαστούμε για να πετύχουμε μια συνένεση και να δούμε ποια είναι τα θέματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για μένα μία από ε, οδούς που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας. Γιατί στη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο, εγώ διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία δεν συμφωνεί με το κείμενο όπως Η τώρα το αρχικό κείμενο. Η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Υπάρχει μια συμφωνία για την απόδοση και την ποιότητα, για την διαφάνεια, ιδίως για το public service obligation, την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών οικουμενικού χαρακτήρα, αλλά το ερώτημα πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κείμενο το οποίο τελικά θα μας επιτρέψει να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Ποιότητα, διαφάνεια, απόδοση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά όπως είπατε γιατί οι επενδύσεις στα συνδεδομικά είναι πολύ σημαντικές και σε οικονομικό επίπεδο και σημαντικές για την κινητικότητα και με τον τρόπο αυτό είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια αγορά για τα σιδηροδρομικά θέματα, αλλά αυτό λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μερών, για μένα είναι σημαντικό και επί τη βάση των ενδιαμέσων εκθέσεων που έχουν γίνει σε διάφορα συμβούλια, μπορούμε λοιπόν επί τη βάση αυτών μπορούμε να φτάσουμε σε μια συνένεση, να τα εγκρίνουμε όλα αυτά τον Οκτώβριο, τι θα κάνουμε μετά. Αν φτάσουμε να έχουμε μια συνένεση τον Οκτώβριο, μπορούμε αμέσως να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους υπόλοιπους πυλώνες που μένουν και εμείς έχουμε δηλώσει όταν αναλάβαμε την Προεδρία ότι θέλουμε να κρατήσουμε τους τρεις πυλώνες την διακυβέρνηση, το PSO και τα τεχνικά θέματα ώστε στο τέλος να ξεκινήσουμε να τα αντιμετωπίζουμε και τα τρία μαζί. Αυτό λοιπόν αφορά το τέλος της Προεδρίας μας και αν δεν καταφέρουμε να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, το ελπίζω και εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξο, τότε θα τα δώσουμε όλα αυτά στους Ολλανδούς οι οποίοι παρακολουθούν πολύ καλά τη συζήτηση και θα μπορέσουν τότε οι κάτω να περατώσουν εργασία αυτή τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο η δική μου ελπίδα είναι όμως ήδη το Δεκέμβριο να έχουμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Με θελησιοκρατία και αισιοδοξία λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει κανείς μια μάχη ούτως ή άλλως. Έρχομαι τώρα στην, στον αεροπορικό κλάδο. Εδώ εμπλέκονται πολιτικά θέματα τα οποία δεν συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με το Συμβούλιο Μεταφορών. Είναι δύσκολα θέματα πολιτικά. Είπατε κύριε Μαρινέσκου ότι έχουμε μια υποχρέωση να προχωρήσουμε σε ένα τριγωνικό διάλογο. Δίκαιο έχετε. Αλλά γνωρίζοντας επίσης τι συμβαίνει, τι έχουμε συζητήσει τους τελευταίους μήνες, τι έγινε κατι τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας, θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν τα εμπόδια. Δεν είναι μοναχα θέμα ενό κράτου μέλου ή δύο κρατών μελών που υπαρχουν τα εμποδια δεν ειναι μοναχα θεμα ενο κρατου μελου η δυο κρατων που μπλοκαρουν την κατάσταση. Είναι μια γενική συγκυρία που δεν είναι πολύ θετική είναι δύσκολη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τουλάχιστον άτυπα να διαπραγματοποιήσουμε διαπραγματεύσεις δίνοντας προτεραιότητα, όπως είπα, στα δικαιώματα των επιβατών γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να το περατώσουμε το ζήτημα αυτό στη διάρκεια της μας. Για τις επενδύσεις, και εγώ καταλαβαίνω τις επικρίσεις σας. Ξέρετε όμως ότι το θέμα της χρηματοδότησης, το θέμα του προϋπολογισμού για τις υποδομές μεταφορών δεν είναι μονάχα θέμα μεταφορών. Είναι κάτι που εμπλέκεται και σε άλλα Συμβούλια Υπουργών και στην Κομισιόν. Μέσα όμως στο Συμβούλιο Μεταφορών η θέση μας είναι ακριβώς στο ίδιο μήκος με αυτά που είπατε. Δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και ημών με ύψιλον. Το μήνυμά σας λοιπόν είναι ένα μήνυμα το οποίο το γνωρίζει το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών για το πόσο σημαντικό είναι το τομέας των μεταφορών και η αρμόδια επίτροπος είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη να υπάρξει μια πρόοδο στο θέμα αυτό. Δεν διαφωνεί καθόλου με το Συμβούλιο. Για τα ποδήλατα, ο κύριος Φανκάπ μου θέτει το αν είσαστε ποδηλάτης. Είμαι ποδηλάτης, μπορώ να σας πω. Κάθε μέρα πάω στο Υπουργείο μου με ποδήλατο για απλό λόγο ότι είναι ο πιο άνετος τρόπος να πάω εκεί. Είναι πολύ απλό. 15 λεπτά ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλα είναι τα ποτηλιάρισμα στο Λουξεμβούργο, εγώ πάω σε 15 λεπτά. Υπάρχουν αυτοί που μου λένε και άμα βρέχει τι γίνεται κτλ. Μα στο Λουξεμβούργο βέβαια δεν έχουμε τον ήλιο του Νότου, αλλά τα καταφέρουμε. Μπορεί κανείς να φορέσει ρούχα βροχής και να κάνει τις διαδρομές που χρειάζεται. Τώρα το αν αξίζει τον κόπο να συζητάμε για τα θέματα της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ή είπε ο κύριος Πίπερ ότι είναι χαμένος κόπος. Έτσι κι αλλιώς θα γίνουν από μόνα τους αυτά τα πράγματα. Για να είμαι σαφής. Δεν είναι η δική μου πρόθεση να ξεκινήσω τώρα συζήτηση για νέους κανόνες για τον τομέα των ποδηλατοδρόμων κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει κανένα νόημα. Μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά στα κρατημέλη, στις περιφέρειες, στις πόλεις. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτός είναι ένας τρόπος μεταφοράς που τον έχουμε υποτιμήσει. Έχουμε υποτιμήσει τον οικονομική σημασία του, όπως είπε και ο Σκράμερ, σημαντική στον τομέα του τουρισμού. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία σε ό,τι αφορά την οικονομική σημασία της ποδηλασίας εν γέννη. Και ξέρουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει αναγέννηση στην ποδηλασία, κυρίως γιατί είναι ένας τρόπος μεταφοράς που προς το παρόν δεν έχει ισοδύναμη σημασία με την, με την ε, πεζοπορία ή με την αυτοκίνηση. Πρέπει να του ξαναδώσουμε τη θέση του και μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προωθήσουμε αυτή την δραστηριότητα χωρίς να θέτουμε κανόνες, αλλά μονάχα με το να δείξουμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που ανοίγονται από τη χρήση του ποδηλάτου. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες λοιπόν για να απαντήσω τώρα σε ένα ερώτημα που έλεγε αν δώσουμε πολλά κίνητρα στις πόλεις με συμφόρηση για περισσότερη χρήση ποδηλάτων. Εντάξει, μα αυτό το ακούμε πάντα, το να, να αυτά τα επιχείρηματα. Θα έλεγα ότι αν δείτε ποιες είναι οι ανάγκες, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα, θέσουμε το, θα να θέσουμε το ερώτημα τι είδους πόλη θέλουμε να έχουμε στο μέλλον. Θέλουμε να έχουμε τις πόλεις που είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιες είναι οι πιο ανταγωνιστικές πόλεις στον κόσμο. Κοιτάξτε τις στατιστικές. Βιέννη, Κοπενχάγη, Βανκούβερ, Μονρεάλ. Είναι πόλεις οι οποίες μπόρεσαν να είναι στην πρωτοπορία για τις νέες μεθόδους κινητικότητας της νέας οργάνωσης του αστικού χώρου και βρίσκονται στο top 10 των ανταγωνιστικών πόλεων στον κόσμο. Κοιτάξτε όλες τις στατιστικές, είναι πάντα οι ίδιες πόλεις. Και ποιες είναι οι πόλεις οι οποίες έχουν τη χαμηλότερη ποιότητα ζωής, τη μεγαλύτερη συμφόρηση κτλ. Αυτό θα πρέπει να δούμε, αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια μέρα. Υπάρχει μεγάλη οικονομική σημασία που πρέπει να συζητηθεί πίσω από τις συμφορήσεις και τα προβλήματα κυκλοφορίας. Δεν πρόκειται να θέσουμε υποχρεωτικούς κανόνες, αλλά πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση. Τέθηκαν και κάποια ερωτήματα πιο συγκεκριμένα. Για τους κανονισμούς σε <clears throat> ευρωπαϊκό επίπεδο, Για το Uber, <clears throat> εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά, <clears throat> αλλά πρέπει να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτό το σύστημα. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα, αυτό είναι σαφές, αλλά τίθενται και κοινωνικά θέματα και φορολογικά θέματα <clears throat> από το σύστημα Uber. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε λοιπόν και υπάρχει ένας παραλληλισμός μεταξύ του Uber και των ερωτημάτων που τέθηκαν σε ό,τι αφορά την, ε, τον αεροπορικό κλάδο. Αν δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε σχέση με ξένες εταιρείες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί αυτές οι εταιρείες μπορούν να λειτουργούν με πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις κλασικές αεροπορικές εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε κατά την άποψή μου το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα του Uber, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι υπάρχει πίσω από το Uber, πρωτού πάρουμε αποφάσεις. Το θέμα των κοινωνικών ζητημάτων στις οδικές μεταφορές. Δεν νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο τη δυνατότητα να υπάρξει μια λύση και δεν υπάρχει και λύση πανάκια η λύση θαυματουργή για να αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια στους δρόμους. Θα πρέπει να δούμε πρώτα ποια είναι η νομοθεσία η οποία ισχύει σήμερα και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτό είναι το βασικό θέμα, αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στην Ευρώπη. <coughs> Κατά τα άλλα, εγώ θέλω να ξεκινήσω μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και γι' αυτό φυσικά ενδιαφέρομαι να ξέρω ποια είναι η άποψη των άλλων κρατών μελών. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε τις θέσεις των κρατών μελών και μετά μονάχα μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Τα ολοκληρωμένα εισιτήρια, τα συνδυασμένα εισιτήρια. Γενικά, η μεταφορές, οι συνδυασμένες μεταφορές ε, θα πρέπει να αυξήσουν το προφίλ τους, να βελτιώσουν το προφίλ τους. Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι μοναχά ο συνδυασμό, αλλά και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ένα σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων που είναι για συνδυασμένε μεταφορές είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζω πολύ. Και προσωπικά ξέροντα ότι δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με την ε, χρήση των εισιτηρίων στα κάτι μέλη και τις τιμέ τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω ότι παρέμεινε και μέσα στο χρονικό διάστημα που μου δώσατε, αλλά ούτως ή ιδάλλως μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε, δεν θα έρθω εδώ μονάχα το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο για να κάνω ένα τελικό απολογισμό. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας αν θέλει το Κοινοβούλιο να συζητήσει κάποιο ειδικό πρόβλημα. Αν έχετε κάποια λοιπόν επιθυμία, πέστε μου και θα έρθω αμέσως. Ευχαριστώ, λέει και ο Και για τα θέματα των προβλημάτων στην Γερμανία που έχουν. Ναι, το θέμα των ε, ελαχίστων αποδοχών των ε, οδηγών των φορτηγών. Ναι, ναι, ναι, ξέρω ότι αυτό είναι, σας είπα ότι είναι δύσκολο να απαντήσω όλα τα ειδικά ερωτήματα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω και η Κομισιόν πρέπει να επιληφθεί για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν είναι η αυτή η οποία υποβάλλει προτάσεις. Δεν μπορεί κανεί να από το Συμβούλιο να το αντιμετωπίσει αυτόνομα. Και σίγουρα αυτό θα είναι κομμάτι και τη συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο. Αν έχει ένα πρόβλημα ένα κράτο μέλος, το οποίο το φέρνει επιτάπητος, σίγουρα πρέπει να συζητηθεί, αλλά εναπόκειται στην Κομισιόν να καταθέσει αντίστοιχε πρωτοβουλίε. Ευχαριστώ και για την τελευταία πληροφορία που μα δώσατε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Μπάου, για την παρουσίασή σα και τι απαντήσει σα. Αυτό το οποίο μα χαροποιεί ιδιαίτερα είναι η αισιοδοξία σα. Χωρί αισιοδοξία δεν πάμε πουθενά και πιστεύω ότι η Λουξεμβουργική Προεδρία μπορεί να έχει τις ευχές μας για το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχω και ηρέμως αν δεν θέλετε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η συγγήτρια είναι η Τζάκλι Φώστα και έτσι είναι το λόγο. Uh, thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προχωρήσουμε λοιπόν. Κάναμε ε, μια περιστατωμένη συζήτηση για το έγγραφο εργασίας πριν από λίγες εβδομάδες και μετά κάναμε και μια σύσκεψη με τους ε, ε, σκιώδης. Ήταν πολύ επικοδομητική η σύσκεψή μας και θέλω να του ευχαριστήσω. Επίσης, έγινε και ε, αρχική συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και τι του είπα και πάλι, ότι επειδή δεν είχε φτάσει το σχέδιο στη μετάφραση προτού να ολοκληρώσουν τη δική τους έκθεση, μπόρεσα να ενσωματώσω σχόλια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στο σχέδιο μου. Οπότε έχω μιλήσει και με τον εισηγητή στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Για όσους δεν ήταν παρόντες θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρόκειται εδώ για την ε, αυξημένη χρήση των μη πανδρομένων ε, οχημάτων. UAS, UAEV, υπάρχουν ε, πολλές και διαφορετικές ορμοθεσίες, αλλά ας λέω drones εγώ γιατί όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Ε, και ε, στο στρατιωτικό τομέα υπάρχει ιστορία δεκαετίων. Το 35 νομίζω ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του Ηνωμένου Βασίλειου για στρατιωτικούς σκοπούς. Ε, με τις εξελίξεις αεροπορίας τώρα φτάνουμε σε αυτό που εγώ αποκαλώ τρίτη φάση. Ε, είχαμε με τα διάφορα αεροπλάνα φτάσαμε στα μη επανδρομένα ε, οχήματα που πλέον δεν είναι ε, κάτι ασυνήθιστο και στον εμπορικό τομέα χρησιμοποιούνται ε, συνήθως αυτά τα drones Τώρα, ε, ήθελα να σας μιλήσω για διάφορες κατηγορίες, αλλά πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει ε, κανένα προηγούμενο εδώ ε, στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τα αυξημένη εμπορική χρήση των drones. Δεν υπάρχει προηγούμενο, δεν μπορώ να παραπέμψω σε κάποια άλλη έκθεση και γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Σίγουρα ε, υπάρχουν πολλά πλέον όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και ανά τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ε, όλοι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στην κατασκευή αυτών των ε, αγαθών. Ε, Καθοριστική σημασία είναι η ρύθμιση της αγοράς ναι. χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς ε, να σταματήσει η εμπορική δραστηριότητα. Αυτό έχει καταλητική σημασία. Λοιπόν, χωρίς να προδικάζω αυτά που, ε, τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε, να σας πω πώς έχει η κατάσταση στον, ε, στην πολιτική αεροπορία. Έχουμε νομοθεσία που θα καλύψει και τα εμπορικά drones, έχουμε και αυτά τα μικρά drones, τα baby Amazon drones, γιατί τα αγοράζουν στο Amazon ή όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, ε, και δεν θέλουμε να σταματήσει αυτή η χρήση επειδή δεν υπάγονται στην, ε, πολιτική, στην πολιτική της πολιτικής αεροπορίας. Ανάμεσα στα δύο υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μη επανδρομένων και τι βλέπουμε τα τελευταία 15 χρόνια και παρατηρείται ημερησίως αύξηση της χρήσης τους είναι ε, για να έλεγχο των συνδρομικών γραμμών, έλεγχο των συγκομιδών, των χωραφιών, ε, για να παρακολουθούν οι αγρότες ε, τις καλλιέργειες, έλεγχος ασφαλείας. Ένας αερομεταφορέας άρχισε να χρησιμοποιεί ντρόνς για να ελέγχει τα αεροσκάφη του παραδείγματος χάρη. Ή εργοστάσια, ή πυρηνικές εγκαταστάσεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ήδη χρησιμοποιούνται και ε, θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς ε, μια κίνηση, γιατί ε, χωρίς όμως να εμποδίσουμε την αύξηση που υπάρχει στην εμπορική χρήση των ε, μη επανδρομένων, έκανα διαβλέψη με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, την κοινωνία των πολιτών, τις αρμόδιες αρχές πολιτικές αεροπορίες, με τις αρμόδιες εθνικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας, κατασκευαστικές εταιρείες, ενώσεις πιλότων, ελεγκτών ερέση κυκλοφορίας. Κάλυψα όλο το φάσμα ε, ε, των εμπλεκομένων φορέων όπου παρατηρείται αντίκτυπος από την αυξανόμενη χρήση των ε, μη επανδρομένων και προκύπτει με σαφήνεια ότι πρέπει με ελαφρύ να αρμοθετήσουμε, δηλαδή να μην υπερβάλλουμε τις οι λεπτομέρειες είναι κάτι που θα αποφασίσουν οι ρυθμιστικές εθνικές αρχές σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει μια δέσμη κανόνων για τους φορείς, για τα ε, μικρά ντρόνους που φτάνουν σε ύψος 400-500 μέτρων. Ε, ε, ο Τζάρος που είναι όπου εκπροσωπείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι κανονιστικέ παντρομένων συστημάτων, έχει μη επανδρομένων συστημάτων, έχει ε, μια επιτροπή που καλύπτει και άλλε χώρε. Οι Αμερικανοί παραδείγματο χάρη συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή και ε, Πρόεδρε, όπω είπαμε και στο παρελθόν, ε, κάναμε μια πολύ υποδομητική συζήτηση με την FAA όταν πήγαμε στην Washington το Φεβρουάριο και είδαμε πώ και εκείνοι θέλουν να το προχωρήσουν το ζήτημα. Νομίζω ότι υιοθετούμε μια ελαφρώ διαφορετική προσέγγιση. Λοιπόν, Επιστρέφοντας τώρα σε αυτό που έλεγα, πρέπει να προσδιορίσουμε πώς ακριβώς θα χειριστούμε το ζήτημα και για να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα θα έλεγα ότι κατά περίπτωση εξετάζουμε τι πρέπει να κάνουμε γιατί είναι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Αν έρχεται ένα ντρόν 150 κιλά και μπορεί να ανέβει με τόση ταχύτητα ε, σε τέτοιο ύψος και σε μία εβδομάδα αλλάξουν αυτά και είναι 50 τα κιλά και άλλα τα μέτρα, το ύψος δηλαδή και η ταχύτητα. Δεν είναι να θέτουμε όρια, τιμές ε, ε, νομίζω ότι οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές ε, μπορούν, επειδή έχουν και τις ε, απαιτούμενες πληροφορίες στη διάθεσή τους, να ρυθμίζουν νομοθετικά ανακατηγορία, ανατύπω πανδρομένου οχήματο και όχι κατά περίπτωση, διότι υπάρχουν πολλοί που μας λένε ότι αν δεν υπάρχει νομοθετική ρυθμίση δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τα κατάλληλα μη επανδρομένα, αλλά αντίθετα, αντίστροφα, λόγω των των τεχνολογικών εξελίξεων θα καταστεί άκυρη οποιαδήποτε υπερβολική νομοθετική ρύθμιση. Αυτά από κατασκευαστική πλευρά. Φυσικά χρειαζόμαστε μια ρύθμιση, χρειαζόμαστε πρότυπα. Έχουμε ε, την, το Ευρωπαϊκό Σήμα σε κάθε περίπτωση και τα αγαθά θα εξάγονται ανά τον κόσμο και θα πρέπει επίση να δεχτούμε ότι αντίστροφα θα εισάγονται ε, και προϊόντα για όσου ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο τώρα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια, η ασφαλής χρήση των μη επανδρομένων και άρα οι χειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ε, επιστοποιητικά αξιοπλοείας ε, από κατασκευαστικής πλευράς. Χρειαζόμαστε επίση στοιχεία για τους ιδιοκτήτες, τους κατόχους. Χρειάζεται αδειοδότηση πιστοποιητικό ε, και επίσης άδεια για τους χειριστές σε μικρότερη κλίμακα, όχι για τα μεγάλα ε, οχήματα και για ε, καταχώρηση αυτών που χειρίζονται παραδείγματος χάρη τα drones. Δηλαδή καταλαβαίνετε όταν είσαστε σε ένα χωράφι όπου καλλιεργείται στάρι δεν θα έχει και πολλούς γύρω γύρω. χρειάζεται καλή κατάρτιση αλλά χειρίζεστε ένα τέτοιο όχημα σε ένα ε, γήπεδο ή σε μια συναυλία ε, με τόσους ανθρώπους ε, τριγύρω θα πρέπει να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι ότι έχει την κατάλληλη κατάσταση και είναι επαγγελματία αυτός που χειρίζεται τον drone και είναι εκπαιδευμένο. Χρειαζόμαστε λοιπόν σχολές για την κατάλληλη κατάρτιση. Πρέπει να φροντίσουμε να είναι καταχωρισμένοι αυτοί που έχουν λάβει την αδειοδότηση για το χειρισμό αυτών των οχημάτων και αυτοί που έχουν την κατάλληλη κατάρτιση θα πρέπει να είναι οι μόνοι που θα μπορούν να χειρίζονται τα οχήματα υπό κατάλληλα προσδιορισμένε συνθήκε. Για μια πυρκαγιά, παραδείγματο χάρη, δεν έχουμε τι ίδιε ανησυχίε για την ασφάλεια γιατί δεν υπάρχει κανένα εκεί. Νομίζω καλύψαμε αυτά τα ζητήματα που έπρεπε, καθώς και το θέμα των δεδομένων ε, και της ιδιωτικής ζωής. Υπάρχει ε, η νομοθεσία για αυτά τα δύο ζητήματα σε εθνικό επίπεδο και ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε αντίστοιχε ρυθμίσεις. Πρέπει να φροντίσουμε μόνο συμμόρφωση, υπάρξει συμμόρφωση σε εθνικό επίπεδο και οι αρχές επιβολής του νόμου να ε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου όταν υπάρχουν παραβιάσεις. Και αυτό είχε συμβεί στο παρελθόν. Έχουμε εμπειρία σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι η κατάσταση ε, προς στιγμή. Ναι. Ε, με τον Νικάου για τα υποπρότυπα έχουμε μια συμφωνία ήδη και είναι εξισορροπημένο το σχέδιο έκθεση κατά τη γνώμη μου. Προσπάθησα να είμαι ε, απλή σαφής, να μην είμαστε ε, υπερβολικά περίπλοκοι γιατί θέλουμε να περάσουμε ξεκάθαρο ε, εναργές μήνυμα προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιθυμούμε να ευθετήσουμε μια διεθνή προσέγγιση και να μην έχουμε υπερβολική νομοθετική ρυθμίση. Αυτά είναι τα δύο μηνύματά μας. Αν θέλουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά και να έχουμε έχουμε έτσι και πρωτοποριακό ρόλο και πλεονέκτημα σε σχέση με άλλου, ε, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, διότι ε, συνειδητοποιούμε όλοι πω με την αυξημένη εμπορική κρίση αυτών των επανδρομένων οχημάτων μπορούμε να έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο όλοι καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστούμε κυρία Κλουμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω εκ μέρου του κ. Μουσουλέγου, ο οποίο είναι ο σχεδόν ηγητή και συμπαθάτε τον. Που δεν βρίσκεται εδώ να σας διαβάσω το σημείο που μου έδωσε. Ε, ελπίζω να σας τα πω σωστά. Πρώτα πρώτα. Ο σκεφτής ευχαριστεί για την έκθεση την κυρία Φώστερ, τη θεωρία αξιόλογη μέχρι τώρα, για τη διάθεσή της, για τις συναντήσεις που είχαν και θεωρεί ότι έχει όλα τα σημαντικά στοιχεία που να βλέπω σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα παρατηρήσεις Πρώτα από το θεωρώ είναι καλή ιδέα να αναφέρουμε και την στρατιωτική χρήση. Όπω είπαμε δεν υπάρχει μόνο η πολιτική χρήση. Προβληματίζεται να μην υπάρχει ε, ε, μην το εκμεταλλευτούν σαν πρόφαση αυτό οι αντίθετοι με τα ε, drones και ε, ε καταφέρουν κατά τρόπο την εμπορική χρήση των μη πανδρομένων σκαφών Λέει ο σχεδόν ότι θα πρέπει σήμερα να επιμείνουμε όσον αφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ασφάλεια των πολιτών. Επίσης το θέμα της ιδιωτικότητας και όσον αφορά αυτά τα ε, μη επανδρομένα σκαφιά διασκέδαση. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα οποία πετούν κάτω από τα 500 πόδια. Ε, όσον αφορά τώρα την πολιτική αεροπλοεία, να πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο ρύθμισης και είπαμε ότι η καλύτερη μακροπνοή είναι να υπάρχει αυτό το 50 κιλών. Επίσης, αγαπημένοι και προβληματίζεται για την δυνατότητα τους να αναλάβουν κάποια καινούργια αποστολή και ας επίσης αν δεν τα καταφέρει πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο, κάποιο άλλο φορέα τώρα για το παράγω 19 θα πρέπει να εξαρτηθούν τα θέματα εκεί να είμαστε πιο συγκεκριμένοι θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι γραφές, αυτές οι προϋποθέσεις θα περιχαρακωθούν καλύτερα. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και εδώ πέρα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε οι πρωτοπόροι σε όλο τον κόσμο, ώστε να έχουμε μια νομοθεσία να εξασφαλίζει ασφάλεια, να είναι φιλόδοξη και όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενεργήσουν και να μην χάσουμε την ευκαιρία. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Ζενκέ, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Φούστα για το εξαίρετο έργο της. Και νομίζω ότι είναι σαφές για όλους μας ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι μονάχα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι και επανδρομένο. Όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε σχέση με αυτό το νομοθέτημα ξέρουν ότι είναι μια περιπέτεια. Μπαίνουμε σε ένα τομέα ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εξερευνηθεί και δεν έχει αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε παρθένο έδαφος βρισκόμαστε. Μετά από την πάρα πολύ λεπτομεριακή έκθεση της ε, κυρίας ε, Φώστερ που διάβασα, δεν έχω καθόλου ερωτήματα επί της ουσίας. Είναι πάρα πολύ ε, λογική αυτή η έκθεση γιατί συνδυάζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη αυτής της μορφής πολιτικής αεροπορίας και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ελληνιστή drones. Ξέρω όμως ότι θα πρέπει να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να ρυθμίσουν τα θέματα των αεροσκαφών αυτών, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν κάνει καμία ε, μέρημνα για τα ζητήματα αυτά. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένας τομέας που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο ενεργή και για ουσιαστικούς λόγους. Μια έλλειψη εναρμόνισης θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούν να πετούν αυτά τα αεροσκάφη από τη μια χώρα στην άλλη. Και θα υπάρξει έτσι μια δυσκολία λόγω έλλειψης ρυθμίσεων ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και αμοιβαία τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας. Για την κυρία Φώστερ λοιπόν θα ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα και να τη ζητήσω να λάβουμε υπόψη και τους κανόνες της ΙΚΑΟ για τα μη ε, επανδρομένα αεροσκάφη. Η ΙΚΑΟ έχει την πιο σημαντική ανάλυση για τα θέματα αυτά, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα σεμινάριο για τα μη επανδρομένα drones και είναι ο μόνος φορέας ο οποίος μπορεί για την πολιτική αεροπορία να θεωρηθεί ότι έχει μία εντολή για να θεσπίσει μία κοινή πολιτική στον τομέα αυτό. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το κεκτημένο της ΙΚΑΟ. Η τρίτη μου παρατήρηση τώρα έχει να κάνει με αυτό το οποίο ανέφερε ήδη η κυρία Φωστέρ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα ότι τα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικό τους σύστημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα drones <clears throat> δεν θα πρέπει να παραδιάζουν αυτήν την νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να συλλέξει κανείς τέτοια δεδομένα, εάν το θέλει κανείς. Θέλω όμως να γίνει μια επισκόπηση των εθνικών κανόνων για να μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσον είναι κατάλληλοι και μπορούν να συναρμοστούν με τη νέα αυτή τεχνολογία και την δυνατότητα να υπάρξει συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων. Το τέταρτο σημείο όμως το οποίο είναι και αυτό εξίσου σημαντικό και είναι το τελευταίο στον κατάλογό μου είναι το εξής. Τι ακριβώς θα πρέπει να διακριβώσουμε είναι το τι είναι νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είναι νόμιμο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίω γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα μηχανήματα με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν αυτά τα ντρόουν θα χρησιμοποιηθούν και για τρομοκρατικές ενέργειες. Πώς μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες. Παράνομες χρήσεις Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε και αυτό το θέμα, λέει ο μιλτής. Ευχαριστώ πολύ. Bilderberg. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα τη δική μου πλευρά και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο την κυρία Φώστερ για την εκθεσή τη. Μας περιγράφει όλο το τοπίο όσον αφορά στα drones. Πάντως, Κατά τη γνώμη μου, Πρόεδρε, θα έπρεπε να σταθούμε περισσότερο στο τι διατάξεις υπάρχουν πέραν του τι συμβαίνει στην πράξη, γιατί θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε γρήγορα, ούτως ώστε να θεσπιστούν κάποιες ξεκάθαρες διατάξεις όσον αφορά το ε, νομοθετικό πακέτο της Κομισιόν. Βλέπουμε εδώ πέρα στο σχέδιο επίση αυτά τα πέντε σημαντικά σημεία. Ε, αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε περισσότερο να φύγουν. πρωτα Πρώτα-πρώτα αυτές οι επιχειρήσεις για τα drones, αυτά θα πρέπει να είναι η αφετηρία για την ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτών των μη παντρεμένων σκαφών. Και οπότε η συνήθι χρήση σε αυτού του είδους την στην επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους. Οπότε πέστε μας κυρία Φώστερ, γιατί μια τέτοια προσέγγιση δεν την επικαλείστε στο κείμενο σας. Δεν είμαι συμπατριώτης σας. Ίσως δεν καταλαβαίνω το βρετανικό χιούμορ. Έχω τέλος πάντων ολλανδικό χιούμορ. Οπότε γι' αυτό σας λέω και σας ερωτώ. Θα πρέπει να αναφερθούμε ε, σε αυτόν τον ευρωπαϊκό οργανισμό και ε, δεν ξέρω αυτό ίσως δεν θα το κάνει κάποιος ε, Βρετανός τώρα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων αναπτύσσονται τεχνολογία για αυτά τα αεροσκάφη αλλά με στην κοινή γνώμη Όμω τι γίνεται, είδατε τι γίνεται το Google Street. Δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τους δρόμους, του ανθρώπου, άρα θα πρέπει και εν προκειμένου να προσέξουμε. Προστασία ιδιωτικότητα, προστασία των δεδομένων. Είναι καθήκον μας. Επίση θα πρέπει να υπάρχει ανεγνευσιμότητα. Θα πρέπει κάπου να καταγράφονται και θα πρέπει να υπάρχει εγκλαισιμότητα του ιδιοκτήτη ο οποίο πάντοτε φέρει ευθύνη για την χρήση του μη παντρομηνού αεροσκάφου. Τέταρτον. Θα πρέπει κανεί να λάβει υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. Να, που θα πρέπει να εμπλακούν οι ρυθμιστικέ αρχέ. Γιατί για όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν όρια, ακόμα και για ένα αεροπλάνο. Τέλος, θα πρέπει να προβληθεί κάποιο κονδύλιο για έρευνα και ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφεύγουμε τα ατυχήματα της συγκρούσεις. Με το geofencing δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα αεροσκάφη αυτά τα οποία πετούν κοντά σε αεροδρόμια ή σε πυρηνικέ εγκαταστάσεις. Προστασία επίση και από του πειρατέ hackers, να μην μπορεί κάποιο να ε, αναλάβει παράνομα την λειτουργία του αεροσκάφου. Οπότε κυρία Φώστα, με όλο το σεβασμό νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές επιδέχονται βελτίωσε. Δεν μπορούμε να πούμε επαναστατικές. Θα συνεργαστούμε μαζί σας όλοι οι σκιώδεις ηγητές. Οπότε θεωρώ ότι όταν ολοκληρωθεί η συνεργασία μας θα μπορέσουμε να εισφέρουμε στο, στο πώς θα ε, εξελιχθεί ε, η πορεία αυτών των ε, αεροσκαφών. Να να δούμε τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. να δούμε το θέμα των αναγκαίων συγγνωτήτων. Θα πρέπει να είναι ασφαλής. Και συμφωνώ τον συνάδελφου. Χρειάζονται κάποια πρότυπα εναρμονισμένα και αυτά να θεσπιστούν ταχαίως. Ε, ε, δεδομένη στις κατάστασεις. Άρα ε, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε αυτό το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειαζόμαστε για την πολιτική χρήση τους, των εσκαφών αυτών, δηλαδή κάποιου κανόνε Οπότε έτσι θα αποκτήσουμε αξιοπιστία. Κατέρινα Κονέσμα έχει το λόγο τώρα. Να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή έχει, την εισηγήτρια έχει καλύψει πάρα πολλά στην έκθεσή της και είναι μια πολύ καλή βάση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον τόσο ενδιαφέροντα τομέα, τον τομέα της χρήσης των drones. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό θα πρέπει να είναι η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων. Πάντα επί τη βάση των εθνικών συνταγμάτων και επί τη βάση του άρθρου της ε, Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του άρθρου 16 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή είναι μια νέα τεχνολογία στον αεροπορικό τομέα. Δεν είναι παιχνιδάκι όπως το λένε κάποιοι κατασκευαστές. Είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις και όσο προχωράει η τεχνολογία και μειώνεται το κόστος κατασκευής, το εργαλείο αυτό γίνεται όλο και πιο προσβάσιμο και όλο και πιο πολύ επικίνδυνο. Όπως και με τα αυτοκίνητα, με τα όπλα ή με τα φάρμακα χρειάζεται να υπάρξει έλεγχος για την λειτουργία τους και την κατασκευή τους. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δει που χρησιμοποιούνται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη για να παρακολουθούν και να φωτογραφίζουν περιοχές οι οποίες κανονικά δεν είναι προσβάσιμες γιατί μπορούν να μπουν σε περιοχές που δεν περιμένει κανείς να είναι υπό παρακολούθηση Για ιδιωτικές γέες, παραγωγός χάρη, υπάρχουν τρόποι να προστατεύει κανείς τον εαυτό του με φράκτες, ώστε να μην είναι ορατές αυτές οι περιοχές. Αλλά αυτό δεν δουλεύει πια με τα drones. Περιμένουμε να υπάρχει πιο πολύ ιδιωτική, ιδιωτικότητα σε χώρους όπως ο δημόσιος χώρος, όπου μας παρακολουθούν συνέχεια οι κάμερες ασφαλείας και είναι ένα άλλο συνδεδεμένο θέμα είναι η ταυτοποίηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και των ιδιοκτητών τους. Δεν ζητώ μεγαλύτερη εναρμόνιση των νόμων για ιδιωτικότητα γιατί νομίζω ότι η τωρινή νομοθεσία στα κάθε μέλη είναι επαρκής. Αλλά, αλλά, αυτό το οποίο θα μπορούσε να τύχει περαιτέρω εναρμόνιση, δύσκολο όσο είναι, είναι ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη των drones εναντίον του οποίου μπορεί κανείς να κάνει αγωγή για παραβίαση ιδιωτικότητας και να ζητήσει αποζημίωση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με το να εγκρίνεται η πώληση στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο ορισμένων drones τα οποία αντιστοιχούν σε ορισμένα τεχνικά πρότυπα. Για, την, για τον εντοπισμό αυτών των αεροσκαφών θα μπορέσουμε ίσως στην αρχή να τα αναγνωρίζουμε με, κάποια, με κάποιο είδος ε, πλάκα κυκλοφορίας για αυτά τα αεροπλάνα τα οποία θα βρίσκονται πάνω στο αεροσκάφος και στη συνέχεια με κάποιο ανέπαφο τρόπο μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Μπορούν λοιπόν έτσι να έρχεται κανείς σε επαφή με τα Μητρώα για την προστασία των προσωπικών ε, στοιχείων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή εφικτό σε οικονομικό επίπεδο για όλους τους ε, χρήστες drones. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αναγνώριση με ειδικέ πλάκες και ε, αναγνωριστικά στοιχεία των ε, drones και μετά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς πομποδέκτες για την αναγνώριση των drones από ένα συγκεκριμένο βάρος η χωρητικότητα τα drones θα πρέπει να καταγράφονται σε μητρό. Αυτό όμως μπορεί όμως να τύχει και περαιτέρω συζήτηση. Και υπάρχει μια άλλη ενδιαφέρουσα λύση που θέλω εγώ να αναφέρω. Είναι η ζώνη μη υπέρπτυσης. Μια περιοχή λοιπόν που η τα drones θα πρέπει να αποφεύγουν και θα βρίσκεται συνέχεια στο λογισμικό των drones. και μόνο τα drones τα οποία σέβονται αυτές τις περιοχές θα μπορούν να την χάνουν έγκριση. Και αυτό ξεπερνάει το πρόβλημα το οποίο είπε, ανέφερε ο συνάδελφος. Κατάχρηση της χρήσεως των drones εκεί που μπορεί να έχουν καταστροφικό χαρακτήρα. Και πάλι αυτή μια πολύ καλή έκθεση για περαιτέρω εργασία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζακή, αλλά παραμένει πολλή εργασία ακόμα μπορούμε να κάνουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι παρά το γεγονό ότι όλοι αποδεχόμαστε ότι αυτά τα drones ήρθαν για να μείνουν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και ανεπαρκής η νομοθεσία μας και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Γεώργιος Βαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Jackie Foster για την τόσο πλήρη και σημαντική της έκθεση αναφέρθηκε σε τόσα πολλά σημεία και ιδίω εξήγησε τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των drones και η οικονομική ε, ανάπτυξη αυτών των ε, ε drones πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλά και η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας για την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση το να υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες και αυτό το χαιρετίζω δεν θέλουμε να παραμείνουμε με ένα καμβά εμβαλωματικό εθνικών ρυθμίσεων. Είναι λοιπόν θετικό να μπορέσει να υπάρξει μια λύση και θεωρώ σημαντικό τα, να υπάρξει ένα όριο των 50 κιλών και να μπορέσει να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση των ευρωπαϊκών drones πέρα από αυτό το όριο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τα ψυχαγωγικά drones. Υπάρχουν πολλές τοπικές περιφερειακές ε, ενώσεις οι οποίες έχουν σαν χόμπι το να πετάνε μοντέλα αεροσκαφών και θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση και για αυτά τα ε, για τον αερομοντελισμό να μην περιλάβουμε και αυτά στον ε, αρμοδιότητες της ΕΑΣΑ. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια σχετική τροπολογία. Αυτό δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε διαμάχες. Όπως σας είπα, πρόκειται για μη ε, εμπορικού χαρακτήρα ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Και γενικά συμφωνώ απόλυτα με την Τζάκι και με την διαδικασία που προτείνει. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει και αυτό την δική του άποψη για αυτήν την ρύθμιση. Κριστίνα Μπουταλόν. Ευχαριστώ. Πρώτα θα ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την εισήγησή τη για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για το μέλλον των αεροπορών για αυτά τα μη παντρεμένα. Για χρόνια ε, από τότε που συνήθω μόνο για στρατιωτικού σκοπού, από τότε υπάρχει τέτοια εξέλιξη, άρα θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη δέσμη για τις αερομεταφορές. Ε, πολλά σωστά έχουμε πει εδώ πέρα. Πρώτα πρέπει να έχουμε ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τι ε, επενδύσει και την απασχόληση στον κλάδο. Τώρα, όσον αφορά και την ε, ασφάλεια, είναι πάρα πολύ σωστό να δούμε πώ θα δώσουμε καινούργιο περιεχόμενο στους κανόνες που υπάρχουν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Ίσως για τα κρατημέλη να δούμε τι θα γίνει που δεν έχουν την αρμόδια αρχή. Οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε φιλελεύθερη προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί η αγορά, ε, αλλά αυτό να μην γίνει βάρο τη της ε, ασφάλειας και ει βάρο τη προστασία τη ιδιωτικότητα, όπω αναφέρεται. Η προστασία των δεδομένων είναι πάρα πολύ βασικό που θα πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητα. Οπότε και οι διάφορε εθνικέ αρχέ να μπορέσουν να συνεργαστούν όσον αφορά τη συλλογή, ε, την διαβίβαση των πληροφοριών, ε, και να υπάρχει σύστημα προστασίας του κόσμου. Οπότε ε, για τα drones αυτά πρέπει να υπάρξει τελικά μέσω του πακέτου ένα πλαίσιο και έτσι να ληφθούν κάποιες αποφάσεις να προωθηθεί ο φάκελο. Ευχαριστούμε Γιάννης Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Κρίνω ότι είναι πάρα πολύ καλό και επίσης ε, αρκετά ευρύ, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων και κάνει μια έκθεση υπεπραγμένων. Χρειαζόμαστε ε, μια δέσμη ευρωπαϊκών ομοιόμορφων κανόνων θα πρέπει να άρουμε το περιορισμό των 150 κιλών μεταξύ άλλων. Χρειαζόμαστε ομοιόμορφη νομοθετική ρύθμιση. Ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια. Δεν ξέρω ποιοι ήταν μαζί μας στον ότι Όταν πήγαμε πριν από λίγες εβδομάδες, ε, μιλούσαμε για τα ντρόνς, ήταν εισηγήτρια φυσικά. Και τώρα τι μας είπαν ότι ε, τα μεγάλα ντρόνς ε, υπάγονται στην ίδια νομοθεσία όπως τα μεγάλα αεροσκάφη ε, και είπαμε ότι χρειάζεται ρύθμιση για τα ενδιάμεσου μεγέθους ε, πανδρομένα οχήματα, όπως σωστά μας είπε η συγγήτρια, ε, όχι για τα μεγάλα και όχι για τα μικρά. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία και ακούσαμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό να έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση. Τα μικρά παιχνίδια, παραδείγματο χάρη, τα παιχνίδια, drones παιχνίδια, δεν μπορούν να φέρουν βόμβες, τι μπορούμε να κάνουμε, να του βάλουμε μια κάμερα και να παρακολουθούμε τι κάνει ο γείτονα. Ε, μέχρι εκεί ε, μπορεί να φτάσουμε. Ε, τίθενται ζητήματα άρα ακαιρεότητας και προσωπική ζωή ακόμη και για τα μικρά επαντρωμένα οχήματα. Θα κατατεθούν τροπολογίες, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το σχέδιο έκθεσης και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε κάποια μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να ξέρει τι θεωρούμε εμεί σημαντικό όταν το φθινόπωρο, ε, πρωτού συγγνώμη, καταθέσει το φθινόπωρο την πρότασή της για το πακέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε και τώρα ο Μάνος Χαρόχια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, Κρατάει υποστήριξή τη ε, σε σχέση με τι προσπάθειε που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νομοθετική ρύθμιση για τα μη επανδρομένα. Έχουμε τα θέματα τη ασφαλεία, ε, ε, τα θέματα περιβάλλοντο και τα θέματα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλα ταυτόχρονα και πώ μπορούμε να προαγάγουμε και ένα ανταγωνιστικό βιομηχανικό περιβάλλον. Επίση, πώ μπορούμε να είναι κανόνε αναλογικοί σε σχέση με τον κίνδυνο, όπω είπατε. Και να προσθέσω και εγώ κάτι, πώ μπορούμε να επιταχύνουμε την νομοθετική διαδικασία, διότι ότι ζητά την σε κανόνε το ταχύτερο δυνατόν. Ε, επεξεργαζόμαστε κανόνες ασφαλείας για τα μη επανδρομένα εχήματα και η ε, πρόταση θα ενταχθεί στο πακέτο αεροναύχειας αεροπλοείας που θα πρέπει να υιοθετηθεί ε, μέχρι το τέλος του 2015. Μετά όμως η ταχύτητα εξαρτάται από τους συνομοθέτες. Ε, ο Άζου θεσπίζει τώρα, η Άζο θεσπίζει λεπτομέρειες τους κανονές ε, για τα μη επανδρομένα εχήματα. Αναφερθήκατε και δύο φορές στον Τζάρους, είναι ένα άλλος αρμόδιος φορέας για τα μη επανδρομένα εχήματα. Ε, και θα, πριν το τέλος του χρόνου και μετά τις θερινές διακοπές ε, θα έχουμε νέες ε, προτάσεις από την ΕΑΖΑ. Χρειάζεται συντονισμός επίσης σε των βιομηχανίας για να εκπονήσουμε ξεκάθαρα πρότυπα. Δηλαδή η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες πληροφορίες σε σχέση με τους στόχους προτού κατασκευάσουν την, τα επανδρομένα οχήματα και φυσικά συνεργαζόμαστε στενά και με τον ΕΑΖΟ και προσπαθούμε να συμβάλλουμε και στην εργασία ε, του ΙΚΑΟ. Ε, επίσης, ε, Αναφερθήκατε κι εσείς σε θέματα ε, ασφάλειας ε, ενσωμάτωσε τη διαχείριση ενέργειας κυκλοφορίας. Ε, εγώ σκέφτομαι δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ε, εντοπισμός του μη επανδρομένου και το geofencing. Είναι η νέα λέξη που έχει γίνει της μόδας και πότε υπάρχει απαγόρευση πτήσης. Όπως είπε και η κυρία Φώστερ, όταν μιλάμε για αερολιμένες, για πυρηνικές εγκαταστάσεις, σημαντικά κυβερνητικά κτίρια, εάν υπάρχει συναρμόνιση για την ταυτότητα ταυτοποίηση των ε, ε, ε, μη επανδρομένων και υιοθετήσουμε μια προσέγγιση geofencing θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια, στην λογοδοσία και στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Έτσι θα μπορούν όλοι εύκολα να ταυτοποιήσουν τα μη επανδρομένα που πετούν γύρω ε, στο τους και θα υπάρχουν και ε, ζώνες απαγόρευσης πτήσης για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τα μία επανδρομένα στις ζώνες διαχείρισης της ενέργειας κυκλοφορίας ε, ζητήσαμε από το ΣΕΖΑΡ την κοινή αυτή τεχνολογική το εργαλείο της κοινή τεχνολογικής ε, πρωτοβουλίας να εξετάσει ε, το ενδεχόμενο ενσωμάτωση των μη επανδρομένων στο master plan της διαχείρισης ε, της ενέργειας κυκλοφορίας ATM και χρειαζόμαστε 40.000 ευρώ για να γίνει μια πρώτη δοκιμή και φυσικά πρέπει να το επανεξετάσουμε τα Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι επιδιώκουμε να βρούμε τεχνικές λύσεις για την αποφυγή των μη επανδρομένων για τα μεγάλα αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά τμήματα εναερίου χώρου από τα μη επανδρομένα και θα υπάρχουν και κοινά τμήματα του εναερίου με τα μεγάλα αεροσκάφη. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε δυνατότητες χρηματοδότησης. Εν κατακλείδη, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Επιτροπή Τρέν και την Εισηγήτρια, διότι είναι εμπεριστατωμένη η έκθεση και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που προσφέρετε. Ε, πολύ θα είμαστε ε, σε στενή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε και πάλι η ε, Τζάκη Φώστερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κομισιόν για αυτά τα οποία ανέφερε. Κατάλαβα ότι έφυγε ο συναδελφός μας από το ΕΛΚ, αλλά θα του τα μεταφέρετε. Ο Δίτερ μίλησε για τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Α, δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα, το διευκρινίζω. Δεν μας ενδιαφέρει η στρατιωτική χρήση των δρόνων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην σφαίρα εφαρμογή του νομοθετήματος αυτού. Χαιρετίζω όμως και πάλι τα σχόλια που έγιναν από το σκιοδησίτη. Έχει απόλυτο δίκιο. Είπε ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτό που λέγεται για τα 150 γραμμάρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παλιωμοδίτικο ως όριο ε, βάρους και εφόσον προχωράει η τεχνολογία δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια τεχνητά όρια. Χαιρετίζω επίσης και αυτά που έχουν να κάνουν με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και από την σοσιαλιστική ομάδα αυτά που είπατε, ναι, είχαμε πολύ καλές συζητήσεις μεταξύ σκιωδών εισηγητών, χαιρετίζω και τα δικά σας σχόλια. Αναφερθήκατε στο όνομα της ΙΚΑΟ. Δεν ξέρω πώς έχει μεταφραστεί αυτό σε διάφορες γλώσσες, αλλά για πολλά από τα σχόλια που έχετε κάνει υπάρχει μία παραπομπή στο βασικό αυτό έγγραφο. Δεν ξέρω αν οι παράγραφοι αντιστοιχούν, αλλά η ΙΚΑΟ ήταν κάτι το οποίο αναφέραμε. Είναι κάτι το οποίο είναι αναπόδραστο και αναπόσπαστο στοιχείο αυτή της πρόταση και, τα θέματα προστασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέραν τα ήδη συνάδελφοι. Πρέπει τα να εφαρμόζουν τους κανόνε τους. Αλλά η δική μου έκκληση ήταν όχι να έχουμε χαλαρότερους κανόνες. Όχι βέβαια, όταν μιλάμε για την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα αλλά να τηρούνται και οι ευρωπαϊκοί νόμοι και οι εθνικοί νόμοι για την ιδιωτικότητα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν πλήρως τι ευθύνες στον τομέα αυτό. Από το Άλδε τώρα. Μιλήσατε και για τον, ε, την ε, ανάλυση επί κινδύνου στην παράγραφο 15. Η ΕΑΣΑ παίζει ένα κομβικό ρόλο στα θέματα αυτά. Είπατε οι αρχε πολιτικη ε, αεροπορια βεβαιω υπάρχουν μερικε εθνικές ε, υπηρεσίες πολιτικη ε, αεροπορια που ασχολούνται με τα, που έχουν κανόνες για τα μικρά μη επανδρομένα τα οποία πετάνε μέχρι 400 πόδια. Η ΕΑΣΑ όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Ερικ Σίβιλ είναι επικεφαλής επιτροπής Γιάρου, ο οποίο είναι ο οποίος είναι στην Επιτροπή αυτή όπου εκπροσωπούνται και οι εθνικοί φορείς. Είναι σαφείς λοιπόν οι αρμοδιότητες και αναφέρονται στην έκθεσή μου. Επίσης σε ό,τι αφορά τα πρότυπα κατασκευής. Και αυτό αναφέρεται στην έκθεσή μου. Και η Κομισιόν αναφέρθηκε στον ορίζοντα 2020 και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Στην πρώτη μου συνάντηση με όλους τους εμπλεκομένους αναφέρθηκα στο ΣΕΖΑΔ, την κοινή σύμπραξη που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα θέματα ενιαίας κυκλοφορίας. Χαίρομαι ότι θα δώσουν και κάποιο χρόνο στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Γενικά, νομίζω ότι έχουν καλυφθεί τα περισσότερα σημεία. Η ασφάλεια φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως είπατε, όταν βλέπετε το θέμα της ασφάλειας, φυσικά δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες ένα μη επανδρομένο μπορεί να είναι μικρό, αλλά πολύ καταστροφικό. Όπως σας είπα, η τεχνολογία προχωρά. Μονάχα τα αεροσκάφη να δείτε και τα ατυχήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ένα σοβαρό ατύχημα μπορεί να είναι και μικρό και όχι κατά ανάγκη μεγάλο. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας που αντιμετωπίζουν αυτό και τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ξέρουμε τι γίνεται και με τις ε, στρατιωτικές περιοχές. Να είσαστε λοιπόν σαφείς για τα θέματα αυτά σε σχέση με την ασφάλεια τα έχω σκεφτεί, αλλά σε επίπεδο διατύπωσης περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει η Κομισιόν για τις λεπτομέρειες. Δεν είναι σωστό εμείς η Επιτροπή μεταφορών να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί εκεί θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές να καθορίσουν τι πρέπει να γίνει τι είδους πρότυπα θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αλλά είπα για όλα αυτά τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οτιδήποτε που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό σήμα, μια πιστοποίηση και να καλύπτονται οι ανάγκες χρηστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν της ταξινόμησης λοιπόν αυτών των αγαθών, είναι απαραίτητο να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, όλα αυτά που είπα λοιπόν και θα συμφωνεί η Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή μόνο μερικά κρατημέρια έχουν κανόνες για τα μικρά μη επανδρομένα. Αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα είναι να περάσουμε σε μια ευρύτερη αντιμετώπιση στην οποία συμμετέχουν πλήρως τα κράτη-μέλη μαζί με την Κομισιόν για να έχουμε απαντήσεις οι οποίες ε, ελπίζω θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ένα πακέτο. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Εάν ξέχασα κάτι, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, αλλά νομίζω είναι απαραίτητο να τα επαναφέρετε αυτά. Εγώ πάντα είμαι στη διάθεσή σας, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και έχουμε κανονίσει μια συνάντηση για τον Σεπτέμβρη. Ραντεβού στο Σεπτέμβριο λοιπόν και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρο. Προθεσμία για 22 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, η ψηφοφορία στις 15 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο αν θέλει ο Θεός. Και για σήμερα το πρωί έχουμε τελειώσει. Στις 3 ώρα το απόγευμα θα επανέλθουμε με τον Pat Cox και τον κόρτο Μπούτριχ. Ευχαριστώ.